Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας, η οποία είναι σημαντική λόγω της ημερησίας διατάξεώς της. Εξού και στο σημείο 1 σχετικά με την υιοθέτηση της ημερησίας διατάξεως να σας, πούμε, να σας πω τις εξής αλλαγές. Το 13 σχετικά με την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Κοστέλο για τη συνοχή αναπτυξιακής πολιτικής ε, για το 2011 θα το συζητήσουμε ε, πριν το 12 όπως προβλέπετε ε, σήμερα δηλαδή πριν την ακρόαση και η κυρία Σρότερ θα προεδρεύσει της Επιτροπής στο σημείο αυτό. Μετά σχετικά με τις ε, ψηφοφορίες για τις γνωμοδοτήσεις η, η έκθεση της κυρίας Μακάρθη ε, για το σημείο 22 και όλα τα σχετικά θα μεταφερθούν για τη συνεδρίαση του Ιουλίου για να ψηφιστούν. Στο σημείο δύο όσον αφορά τα πρακτικά μπορείτε να μου στείλετε τα σχόλιά σας μέσω διαδικτύου και τώρα στο σημείο τρίτη δίνω το λόγο στη κυρία Στάινρουκ για να μας πει ποια είναι η τοποθέτησή της σχετικά με ε, τις ε, τροπολογίες ε, τις συμβιβαστικές μάλιστα τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές ήταν εξαιρετική. Όλοι εργάστηκαν σκληρά συναντηθήκαμε τουλάχιστον 10 φορές και από κοινού εκπονήσαμε τις θέσεις μας και ελπίζω ότι θα έχουμε ένα ευρύ πλαίσιο όσον αφορά τις τροπολογίες και μέχρι το τέλος υπάρχουν ακόμη ορισμένες εκκρεμότητες Ελπίζω όμως ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ θετικό. Παραδείγματο χάρη, αυτό το οποίο βελτιώσαμε είναι ότι έχουμε κατακρίνει ότι η ε, Επιτροπή δεν έχει ε, κάνει ένα κοινό πλαίσιο και το άλλο το οποίο ε, συζητήσαμε είναι ένα κοινωνικό πλαίσιο για καλή απασχόληση, να έχουμε ένα στρατηγικό όργανο διαβουλεύσεων που θα, συμμετέχουν, θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα δεσμευτούν ε, στην αξιολόγηση του, προ... προγράμματος μετά ε, όσον αφορά το συνολικό ο πρόγραμμα το διευρύναμε ε, αλλά ε, ε, έχουμε κατευθυνθεί βάσει της, των υποδείξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κοινωνικές με το κοινωνικό επιχειρήν, τα κοινωνικά πειράματα, τους κοινωνικούς στόχους και πρέπει να διευκρινίζουμε γιατί δαπανά ο καταναλωτής ε, και φορολογούμενος τη συνδρομή του και πού θα καταβληθούν το 1 ε, δισεκατομμύριο ευρώ. Ε, επίσης, ε, αν πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό επίπεδο διαβίωσης ε, ή εάν θα καταλήξουμε σε ένα κοινωνικό παρανομαστή και από κοινού θα μπορέσουμε να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες. Σε κάθε άξονα χρησιμοποιήσαμε τις τα στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και χαίρομαι ιδιαιτέρως να μπορέσουμε όλοι να δημιουργήσουμε ένα νέο άξονα επί του οποίου θα καταπολεμήσουμε την ανεργία και ελπίζουμε ότι αν όντως ε, το Συμβούλιο είναι σοβαρό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, βρούμε πόρους για αυτόν τον κοινωνικό στόχο που θα ισχύσει μόνο εάν προσθεθούν και επιπρόσθετοι πόροι τους οποίους θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε σχετικά με την κοινωνία των πολιτών θελήσαμε να περιλάβουμε το πρότυπο του ESF εις το πρόγραμμά μας και να υπάρχει ένα στρατηγικό όργανο διαβουλεύσεων. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα μας, είναι μία ένδειξη για το μέλλον των ε, διασυνοριακών συνεργασιών που είναι ένας άξονας του προγράμματός μας και θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν διότι αυτό μας το αποδεικνύουν και όλες οι ενδείξεις από τα κράτη-μέλη όπου μας ε, λέγεται ότι δεν θα υπάρξει πλέον χρηματοδότηση μέσω του ESF. Ελπίζω ότι αυτό θα στηριχτεί από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα μπορέσει να υπάρξει μία καλύτερη επάνδρωση του προγράμματος κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να έχουμε και άλλους πόρους πέραν των αρχικών. Ε, έχουμε ένα πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριμένο τώρα από ότι ήταν το αρχικό της διατύπωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε διάφορα θέματα και θέλω να ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία καθότι όλοι εργάστηκαν σκληρά. Τους ευχαριστώ όλους και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε ε, μία θετική έκβαση και ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη σοβαρή παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπλό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της ε, εργασία την οποία επέβλεψε. Ευχαριστώ και τους Κεώδης. Οι συζητήσεις ήταν ε, πλούσιες και επικοδομητικές ε, υπήρξαν πολλοί συμβιβασμοί. Συμφωνούμε με τα πολλά σημεία που ανέφερε. Εμείς επισημαίνουμε την τοπική απασχόληση και η κινητικότητα στο τρέχον πλαίσιο δεν μας φαίνεται προτεραιότητα. Υπάρχουν τα διασυνοριακά ζητήματα και ο άξονας γιορές. Θελήσαμε να επισημάνουμε περισσότερο το progress και τη μικροχρηματοδότηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας όσον αφορά την εγχώρηση ποσοστών που συζητήσαμε. Παραμένει αναρρύθμιστο σημείο που θα συζητήσουμε με το ΕΛΚ σήμερα το απόγευμα και αφορά το ποσό του 5% που Θέλουμε να μειώσουμε ε, κατά 2% και το 3% που θα έμενε στο ΕΛΚ έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε στη μικροχρηματοδότηση. Θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει πραγματικό πρόβλημα όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Εμείς θα τις υποστηρίξουμε κατά προτεραιότητα με αυτό το 3% αλλά δεν μπορώ να προκαταβάλω την αποφάση του ΕΛΚ. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ολοκληρωμένο, στο οποίο έχει προσθέσει την καινοτομία για τους νέους. Φαίνεται να είναι μια καλή απάντηση για τα προβλήματα απασχόλησης του σήμερα. Όσον αφορά την κοινοτομία και τις κοινωνικές αλλαγές, ε, ευχαριστώ την εισηγήτρια που δέχθηκε τις λίγο πρωτότυπες ε, προτάσεις μας που ελπίζω να είναι επικοδομητικές και να βοηθήσουν στην πρόοδο και στην κοινωνική σύγκληση στα πιλωτικά προγράμματα που έχουμε παρουσιάσει. Η κυρία Αρκίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα, οι ειλικρινές ευχαριστίες προς τον εισηγητή πάντοτε, πάντοτε λέμε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τις και όδες και συνήθως το λένε και έχουν δίκιο, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση έκανε τεράστια προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις για να μπορέσει να συγκεντρώσει μια συνένεση. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε, έχουμε μόνο κάποια λεπτομέρειε μόνο να συζητήσουμε, δεν θέλω να μπω τώρα στι λεπτομέρειε, το έκανε η εισηγήτρια. Ε, και απλώ θα σα θίξω πώ να τα συζητήσω. Αλλά επαναλαμβάνω κατά 99% είμαστε ικανοποιημένοι. Στην τροπολογία υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με ε, το φορολογικό και την ισότητα των φίλων. Πρέπει να το δούμε. Επίση, στην τροπολογία S, λατινικό, σε σχέση με την κρίση, ρυθμίστηκε ένα θέμα που υπήρχε με συμβαστική τροπολογία. Ε, γιατί να το θυμάμαι αυτό το πρώτο που υπάρχει η κρίση και μέχρι πότε θα διαρκέσει την Πασχόλη 2016-2017. Θα δούμε τώρα επίση για την κοινωνική διακυβέρνηση. Αυτό είναι ένας νέος όρος και ο κύριος Μπουλόν ε, ξέρω ότι αγωνιά να εμφανιστεί αυτό στην έκθεση σύμφωνη. Εντάξει, αλλά να δούμε τι θα γίνει με την σημαντική τροπολογία ε, γιατί την καθιαυτή διάταξη θα την καταψηφίσουμε τώρα στο Q, στην τροπολογία Q. Εκεί αναφέρεται το δικαίωμα των εργαζομένων και θεωρούμε ότι θα πρέπει να μιλούμε για αυτά σε επίπεδο ένωσης και όχι τα δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το καταψηφίσουμε, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα αποτελούσε πιο εύστοχη διατύπωση. Και το τελευταίο σημείο είναι... Α, Το LLL. Και σε αυτό το σημείο δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη, μεγάλη απαρίθμηση. Ας πούμε εκεί που λέγεται τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας. Είμαι υπέρ της κοινωνικής οικονομίας, αλλά με απασχολεί το ότι έχουμε τόσο λίγη χρηματοδότηση που θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες οι ενεργείες μας. Και έχουμε εδώ πέρα έναν πάρα πολύ μακρύ κατάλογο. Και άρα θα έχουμε διαδιασπάθηση, θα έχουμε ε, σκόρπισμα αυτών των, των χρημάτων. Επομένως, για όλα τα άλλα που σας είπα εκτός από το θέμα το δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Συγχαρητήρια πάλι στην εισηγήτρια. Πολύ καλή έκθεση. Πρόεδρος. Κυρία Ντελή. Συγγνώμη κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Στάινμπρουκ για την ποιότητα της εργασίας που μας παρέδωσε και τις συνεργασίας, της που είχαμε με όλους τους συνεισηγητές, εξαιρετική συνεργασία σε όλη τη διάρκεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. όσον αφορά την τεράστια προσπάθεια συμβιβασμών καταλήξαμε σε συμβιβασμούς και αναδεικνύει αυτό το πρόγραμμα την τεράστια πρόκληση της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας που αναδεικνύουμε σε αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζοντας τους κοινωνικούς εταίρους και τις δραστηριότητές τους και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ενισχύοντας τον κοινωνικό πειραματισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που ήθελα να πω επίσης, ναι, αληθεύει ότι το να βρούμε ορισμούς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τα λοιπά ήταν δύσκολο. Πιστεύω ότι οι σημερινοί συμβιβασμοί μας ικανοποιούν. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας ε, ε, αυτή την πολιτική ε, καινοτομία και αυτή την συλλογική ευφυΐα για αυτό τον τέταρτο πυλώνα που αφιερώνεται κυρίως στην νεολαία. Θεωρώ, ότι πρέπει να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε αυτή την τυχή δεδομένου ότι η κατάσταση των νέων όπως βλέπουμε σχεδόν παντού στην Ευρώπη είναι δύσκολη, δυσκερής και οι νέοι χρειάζονται το κοινοβούλιο μας ώστε να τους ενθαρρύνει, να τους καλέσει να συμμετέχουν σε, καινοτομίες, σε πρωτοβουλίες καινοτομίας. Καλό είναι λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε έναν πυλώνα ώστε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και να διασφαλίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό απασχόλησης, ε, ε, μια εγγύηση υλοποίηση του ευρωπαϊκού ονείρου, οράματος. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και την κυρία συγγήτρια η κυρία Τσίμερ και μετά ο κύριος Τόμας Μάνου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να υποφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω την κυρία Σάινρου και τη θαυμάσια εργασία την οποία έκανε ε, διότι υπήρχαν 92 192 ε, τροπολογίες εκ των οποίων έχουμε 125 δηλαδή είναι ε, η πρώτη προσπάθεια καταρτήσεως εκθέσεως από την κυρία Στάινρου και τη συγχαίρω διότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό και όσον αφορά αυτά που είχε παραλείψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να υπάρχει στην πρόταση μία σωστή δομή και ένα συγκεκριμένο στόχος, τονίστηκαν από αυτή τη γνωμοδότηση και έτσι περαιτέρω μπορούμε να προχωρήσουμε πιο επικοδομητικά. Η πολιτική μου ομάδα σε πολλές ε, ε, τροπολογίες ε, συμβιβαστικές παρόλο που δεν τις έχει συντάξει θα τις στηρίξει και στη συζήτηση αυτή πρόκειται για το κοινωνικό επιχειρήν. Ως εκ τούτου θα σκεφτούμε ακριβώς πόσο θα συμπεριφερθούμε σε κάθε τροπολογία ή σε κάθε συμβιβαστική. Ε, θεωρούμε ότι η συζήτηση και ε, η εξέταση του θέματος του κοινωνικού επιχειρήν είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι το σχέδιο το οποίο απλώς παρουσιάζει παρουσίαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι οι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούνται σαν ένα τομέας μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων με το οποίο δεν συμφωνούμε και γι' αυτό χαιρόμαστε ε, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που έχει προτείνει η συγγήτρια και ως εκ τούτου θέλω να ευχαριστήσω περαιτέρω διότι όσον αφορά την διασυνοριακή δηλαδή κινητικότητα. Οι ε, τροπολογίες ε, έχουν ε, υιοθετηθεί και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως και οι συνεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα πρέπει να προωθηθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία Στρέτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι ότι υπήρξε τόσο ευρία συνένεση για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Δεν πρόκειται απλούστατα για μία νομοθεσία επί της οποίας κάνουμε ένα ψήφισμα ή μία αιτιολογική έκθεση απλούστατα. Θελήσαμε να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά ότι θα ίσχυαν ε, οι αρχές που πρεσβεύουμε. Σχετικά με αυτά που είπε τώρα η Μέρι Χάρκινγκ, δηλαδή την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Είναι να μην λέμε απλώς ε, θέλουμε να είσαστε παρόντες αλλά θέλουμε να σας ε, χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά να έχουμε επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους και με άλλες κοινωνικές οργανώσεις διότι διαφορετικά δεν θα είχαμε μία συνεχή συνεργασία δεν θα υπήρχε ο συνεχής αυτός ε, διάλογος και γι' αυτό θεωρούμε τη διατύπωση πολύ θετική. Επίσης πολλές οργανώσεις οργανώσεις δεν μας συμπαθούν ε, εμάς τους βουλευτές ή δεν έχουμε επαφές και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει τριμερής διάλογος όσον αφορά την ανεργία των νέων όχι απλώς να ε, έχουμε άδεια λόγια αλλά ουσιαστικά να αποδεσμεύσει πόρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο ότι χρειάζεται νέα χρηματοδότηση απλούστατα θα πρέπει να καταρτιστούν τα βασικά θέματα και αυτά να γίνουν σεβαστά δηλαδή ε, δεν υπάρχει αντίρρηση. Ε, ε, ε, δεν χρειάζεται να λέμε απλώς ότι οι νέοι είναι μια χαμένη γενιά. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Επίσης αυτό που είπε ο συνάδελφος ότι στο ΕΛΚ θα το ξανασυζητήσουμε διότι το ΟΗΡΟΣ είναι μια πολύ σημαντική συνεργασία διασυνοριακή η οποία πρέπει να προσδώσουν μια επιπρόσθετη αξία εις το σύνολο. Υπάρχουν αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κονδύλι στον προϋπολογισμό και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει αυτή η διασυνοριακή συνεργασία στα πλαίσια του Εύρος και εάν δεν, επιτρεφτεί, δεν επιτραπεί τότε ε, θα θεθεί σε κίνδυνο μία αρχή την οποία έχουμε θεσπίσει και αυτό πρέπει να αποφευθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι αύριο θα υπάρξει ευρεία συνένεση και το ότι υπάρχουν τόσες πολλές ε, τροπολογίες αποδεικνύει ότι όλες οι πολιτικές ομάδες το εξέτασαν πάρα πολύ προσεκτικά και θετικά και γι' αυτό ελπίζω ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν και αύριο κατά την ψηφοφορία. Πω, πω, πω. Βλέπω ότι ε, ήσασταν πάρα πολύ θετικός για την εισηγήτρια. Η κυρία Σρότερ, πρέπει και εγώ να σας πω ότι αυτή η διαδικασία ήταν πολύ επικοδομητική και ε, ε, το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Άλλο είναι να ψηφίζουμε κατά συρροή 300 τροπολογίες ή εάν υπάρχουν αν υπήρξαν συνεκτικές συναντήσεις που κατέληξαν σε λογικές ε, τροπολογίες ε, κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσει κανείς να έχει μία σωστή συνεργασία στην Επιτροπή όπου όλοι συνέβαλαν, παρουσίασαν τις προτάσεις τους και αυτό για τις διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντικό διότι ξέρετε ότι είναι στα πλαίσια του MFF και έχουμε μία σαφή θέση ε, σχετικά με τις ανάγκες των ε, πολιτών ε, στην Ευρώπη και ιδίως στην ανεργία των νέων. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην συνεργασία στα πλαίσια του Εύρος ε, θεωρώ ότι οι συνεργασίες αυτές οι διασυνοριακές είναι πολύ σημαντικές. Βέβαια ο επιβάρυναν το απόθεμα και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία παρακολούθηση της τρέχουσας ε, ε, διαδικασίας και σαν ευρωβουλευτές να παρακολουθήσουμε πώς κατανείμονται οι πόροι. Ένα θέμα με το οποίο δεν συμφωνούμε είναι το σημείο όπου λέγεται ότι δεν χρειάζεται ορισμός για την κοινωνική καινοτομία διότι εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνική καινοτομία είναι ένας πειραματικός τομέας και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό. Όλες οι άλλες βασικές ε, ε, προϋποθέσεις, ε, ποιος θα χρηματοδοτηθεί, ποια είναι τα βασικά σημεία, όλα αυτά είναι καλά. Βεβαίως τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο στόχο. Αλλά ένα μέσο για την καινοτομία να περιοριστεί να το περιορίσουμε με το, την απουσία ενός ορισμού του τι είναι δεν νομίζω ότι είναι σωστό και δεν θα μπορέσουμε να επαγρυπνήσουμε σωστά εάν δεν υπάρχει αυτός ο ορισμός. Ε, υπάρχει μία προσθήκη που χρειάζεται εδώ και εγώ ε, έχω επιφυλάξεις αν θέλουμε να προχωρήσουμε επί της οδού αυτής. Κυρία Εστρέλα, πρώτη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με εκείνους οι οποίοι συνεχάριζαν την εισηγήτρια. Ήταν άριστη η προσπάθεια που έκανα και έχουμε βέβαια ένα σωρό τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και μία σειρά από συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στις ε, τροπολογίες τη Επιτροπής Γυναικών. Νομίζω ότι πρέπει να, βρει, να βρουν σύμφωνη την εισηγήτρια αλλά και την Επιτροπή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσαρμόσει την νομοθεσία της στις ανάγκες της ε, εποχής. Χρειάζεται ευθύς νομοθεσία. Χρειάζονται εξελικτικές μορφές εργασίας και να αντιμετωπίσουμε τους νέους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια τους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε θα πρέπει να συγκεράσουμε να συμφιλώσουμε την επαγγελματική με την ιδιωτική οικογενειακή ζωή και για τους άντρες ισχύει αυτό και για τις γυναίκες. Επίσης, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να γίνει ελαστικό το ωράριο εργασίας και να υποστηρίξουμε έτσι τον οικογενειακό βίο. Έτσι, να δούμε πώς θα υπάρχουν περισσότερες γονικές άδειες για τον πατέρα και για τη μητέρα. Και επίσης θα πρέπει να διευκολύνουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες. Και έτσι να έχουν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις. Να έχουν περισσότερη επομένω απασχολησιμότητα για τις γυναίκες. Να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους του προγράμματος Ευρώπη 2020. Το 2010 θεσπίσαμε αυτή τη μικροχρηματοδότηση και έτσι θεωρήσαμε ότι βοηθάμε την απασχολησιμότητα. Έτσι επίσης καταπολεμούμε την φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που να λάβουμε υπόψη επομένω και αυτή την διάσταση Τη ισότητα των φύλων στην λόγω έκθεση. Να λέμε υπόψη το πρόγραμμα για, την, για, την, ε, για τις κοινωνικές μεταβολές. Ε, Πάντω σίγουρο ότι μπορούν πολλά να κάνουν γυναίκε όσον αφορά την προσαρμογή μα στη σημερινή πραγματικότητα. Κυρία Σανκλέρ και μετά κυρία Μακεντάιρ. Ε, ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την συγγήτρια για τη σκληρή δουλειά που αφιέρωσε σε αυτή την έκθεση. Μπορεί να μην συμφωνώ με ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά αναγνωρίζω το σκληρό της έργο. Αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά για το Ηνωμένο Βασίλειο και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα, όπως το βλέπω εγώ, είναι η υλοποίηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαδοχικές μας ε, κυβερνήσεις και διάφορες ε, δημόσιες υπηρεσίες έχουν εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πολύ πιο αυστηρά από ό,τι οι εταιρεία μας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε χρησιμοποιήσει τον όρο gold plating γι' αυτό και έχω παρατηρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν έχει κανένα μηχανισμό ώστε να φέρει ε, στο επίπεδο του υλοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό γίνεται εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας και θέσεων εργασίας. Ελάχιστη είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μικροπιστώσεις, αλλά η δική μας κυβέρνηση φαίνεται να εμπλέκεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να υποστηρίζει τους Βρετανούς εργαζομένους. Εδώ έχουμε δύο εκπροσώπους, Μπένιαν και Μακεντάιρ, που είναι βουλευτές της κυβέρνησης και κανείς δεν λέει ότι θα υποστηρίξω περισσότερο τη θέση της κυβέρνησής μας. Ε, μάλλον κρύβονται πίσω από τις ασφαλείς της ομάδας τους. Ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύω, έχει δεχθεί αυστηρές έχει επικρίνει σοβαρά αυτή την έκθεση, ειδικότερα τον αυξημένο προπολογισμό σε εποχέ λιτότητας και πάλι αυτό το κοινοβούλιο είναι το ίδρυμα που δεν γνωρίζει το πραγματικό νόημα της λιτότητα, δίνει μαθήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λιτότητα, αλλά αυξάνει του προπολογισμού σε κάθε επιτροπή Οπουδήποτε βρίσκομαι βλέπω σημαντικές αυξήσεις ε, προϋπολογισμού ενώ ζητάμε από τους άλλους να μειώσουν τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να εφαρμόζετε αυτά που διδάσκεται. Η, αλλαγή, η εφαρμογή των κανόνων σας, ε, η έλλειψη ε, εκτίμησης αντικτύπου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ξέρετε πόσα email λαμβάνω κάθε μέρα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μου λένε σας παρακαλούμε σταματήστε τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας στραγγαλίζει, μας διώχνει από την αγορά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που παράγει αυτό το μέρος μας κοστίζει. Και σε άλλες χώρες φυσικά και στην Ιρλανδία πρόσφατα άκουσα το ίδιο και το, άκουσα το ίδιο από Ιρλανδούς. Έχουν βαρεθεί την έλλειψη κατανόησης των συνεπειών των δικών σας κανόνων και υλοποιήσεων στη δική τους οικονομία και στις θέσεις εργασίας τους. Η ε, κυρία Μακιντάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας διαβεβαιώ ούτε ο κύριος Κάμερον ούτε ο κύριος Κλέγκ υπολογίζουν στην βοήθεια, στη στήριξη από την κυρία Σενκλέρ. Τα περισσότερα από αυτά που είπε αφορούν το επόμενο θέμα τη στη διαταξή, όχι το τώρα συζητούμενο, τέλο πάντων. Για να συζητήσουμε για το θέμα μα. να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο τη. να έχουμε ούτω ή υπήν τροπολογίε. θα βοηθήσουν, ε, μπράβο της, η δική μα ε, πολιτική ομάδα, θεωρεί θετικέ προτάσει επιτροπή. να έχουμε έτσι μια συνέχιση των ισχυών των προγραμμάτων και επίσης να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις προτάσεις όσον αφορά τις δράσεις για κοινωνική καινοτομία και πειραματισμό, έχουμε επομένως με αυτόν τον τρόπο ε, ανταλλαγή των ορισμών πρακτικών και η αλήθεια είναι ότι δεν κατεβάσαμε από αυτού ε, τροπολογίες έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες να σας πω ότι βλέπω διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψηφίσουμε μια αύξηση του προπολογισμού. Ε, το θέμα δεν είναι να ξοδεύσουμε περισσότερα, να ξοδεύσουμε λιγότερα και πιο αποτελεσματικά. Επίσης μας προβληματίζουν ε, διάφορα σημεία ε, επί των οποίων συμφωνούμε για τις καλές προθέσεις, αλλά θεωρούμε ότι αυτές οι δράσεις που προτείνονται αποτελούν επικάλυψη ισχυουσών πράξεων και προγραμμάτων. Και έτσι θα καταλήξουμε να ανταγωνιζόμεθα τις ε, υπηρεσίες προνοίας των κρατών μελών. Επίσης, μας προβληματίζει αυτή, αυτή η τέταρτη δράση πρόσβαση των νέων. Εντάξει, ναι, θα πρέπει κάπως να βοηθήσουμε τα νέων, αλλά να δούμε τι γίνεται με την οριζόντια αγορά εργασία και όχι ε, τομεακά και να κάνουμε τέλο πάντων καλύτερη χρήση των πόρων. Έχουμε ένα σωρό επίσης ε, τροπολογίε, συμβαστικέ, όπως και με τη μικροχρηματοδότηση, με τα οποία συμφωνούμε και νομίζω οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε είναι υπέρ. πάντω θα ήθελα να σα τονίσω ποια είναι η θέση τη πολιτική μα. ομάδα. Και πάλι ευχαριστούμε την συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο ξανά στην εισηγήτρια. Σας ξαναδίνω το λόγο και μετά θα προσθέσω δύο σημεία που θέλω να αναφέρω. Ευχαριστώ. Καταρχήν χαίρομαι ε, ότι ε, επενέθηκα αλλά παραπέμπω του επένους ε, για όσους συνεργάστηκαν με την εισηγήτρια, την γραμματεία και όλους τους άλλους γιατί η εργασία αυτή κατανεμήθηκε και χαίρομαι και συμμετέχω σε αυτόν τον έπαινο αλλά όχι στις κριτικές οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συζήτηση γιατί όσοι συμμετείχαν αν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι προσπαθήσαμε να εξετάσουμε σοβαρά ώρες τις παρατηρήσεις ε, και στην συζήτηση ε, εκφράστηκαν απόψεις προς όλες τις κατευθύνσεις και γι' αυτό βλέπω ότι ορισμένες πολιτικές ομάδες έχουν ε, διατυπώσει κριτικές χωρίς καν να κάνουν την προσπάθεια να υπάρξει μία θετική πολιτική ε, διατύπωση και βλέπω ότι όλες οι απόψεις αντικατοπτρίζονται εις ε, την γνωμοδότησή μας όπως παραδείγματο χάρη είναι οι θέσεις ε, της ε, Επιτροπής Γυναικών για το πρόγραμμα προόδου σχετικά με τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες. Πολλές φορές έχουμε τονίσει στη γνωμοδότησή μας ότι η διευκρίνηση και η αποφυγή διακρίσεων πρέπει να παραμείνουν στόχοι του προγράμματός μας. Εδώ θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι εάν θέλουμε να μειωθεί η ανεργία των νέων, νομίζω ότι ο καθένας ο οποίος πιστεύει ότι χωρίς ε, συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένες ε, καινοτομίε στην Ευρώπη αυτό δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί και γι' αυτό περιμένουμε τα νέα προγράμματα. Ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση είναι στενάχωρη. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά που βρισκόμαστε στην Ευρώπη και πώς πάνε τα οικονομικά μας. Γι' αυτό όμως πρέπει να δώσουμε μία ένδειξη καθότι μιλάμε εδώ και χρόνια για την μείωση της ε, ανεργίας των νέων χωρίς να συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο και αυτό το αποδεικνύουν και οι αριθμοί. Έχουμε περιλάβει και ε, ορισμούς γιατί έπρεπε να διευκρινίσουμε ε, πού διατίθενται τα χρήματα και εάν ε, συζητάμε για το θέμα της, ε, του κοινωνικού επιχειρήν ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται δεν πρέπει να εμπλέκονται. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε πολύ πώς θα, ε, θα διαμορφωθεί τελικά η διατύπωση. Θέλω επίσης να πω σε όλους ότι έχουμε καταλήξει σε συμβιβαστικές τροπολογίες για τη διασυνοριακή συνεργασία και της ε, ε, ε, η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΟΡΟΣ δεν έχει αφαιρεθεί από άλλο πρόγραμμα αλλά τονίζοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση χρηματοδοτήσεως σε άλλα προγράμματα που μας απασχολούν. Αλλά πιστεύω ότι ήταν επιτυχής η συμβιβαστική και τροπολογίες και γενικώ η συζήτηση ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις τους. Προσπαθήσαμε ε, με συγκεκριμένες θέσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τελικά κάπως τα καταφέραμε και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγήτρια. Θα ψηφίσουμε για το κείμενό σας αύριο. Εγώ ήθελα να δώσω τρία μηνύματα. Το πρώτο που αφορά αυτή την ψηφοφορία για την οποία χρειάζομαι φυσικά και την άποψη των συντονιστών και επίσης για δύο άλλες πτυχές που αφορούν την έκθεση. Το πρώτο στοιχείο θα θυμάστε όταν θα ψηφίσουμε αύριο για αυτή την ε, γνωμοδότηση θα αποτελέσει την πρώτη νομοθετική βάση βάση της οποίας θα ε, ψηφίσει μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Είμαστε οι πρώτοι. Δεν ξέρω αν είμαστε πειραματόζωα, αλλά είμαστε οι πρώτοι. Έτσι λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόζουμε τον κοινό κανόνα που έχει εφαρμοστεί ότι στις νομοθετικές βάσεις δεν προκαταβάλουμε την τελική συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπήρχαν αριθμοί υπάρχουν τώρα παρενθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν αριθμοί και ότι αν οι τροπολογίες δεν περιλαμβάνονται στους συμβιβασμούς και περιλαμβάνουν αριθμούς δεν θα ψηφιστούν. Σας υπενθυμίζω αυτόν τον κανόνα και θα σας τον υπενθυμίσω και αύριο ώστε να μην υπάρχουν εκπλήξεις και με να αρχίσει να λέω καθένα, ναι, δεν ψηφίστηκε η δική μου τροπολογία. Εάν περιλαμβάνει αριθμού, μεγέθη, δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία. Το δεύτερο, όσον αφορά τη γοητεία των πρώτων αναγνώσεων και των διαπραγματεύσεων, ε, είμαστε λίγο σε δύσκολη θέση, διότι η πρακτική μας, που πιστεύουμε αντιστοιχεί στην πρακτική του Κοινοβουλίου, είναι να, ξεκινά, να κάνουμε διαπραγματεύσεις ε, βάσει της εντολής που μας δίνει η Επιτροπή Απασχόλησης και να προσαρμόζουμε την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια εντάσσοντας για την Ολομέλεια τις τροπολογίες που επιτρέπουν να λαμβάνουμε υπόψη τους συμβιβασμούς που έχουν μελετηθεί μαζί με το Συμβούλιο πριν καταλήξουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Είναι μια πρακτική που μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει καλά μία από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου με την οποία συνεργαζόμαστε στενά επιθυμούσε να ξεκινήσουμε μια άλλη διαδικασία η οποία θα συνίστατο στη ψηφοφορία των τροπολογιών αλλά στο να μην γίνει τελική ψηφοφορία του κειμένου. Όταν συνεδριάσαμε ως ομάδα επαφής χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανέφερα αυτό το ζήτημα, μας ζήτησε να αναβάλουμε οποιαδήποτε ψηφοφορία πριν αυτό το ζήτημα ρυθμιστεί σε όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα, ωστόσο, έχουμε λάβει εντολή να προχωρήσουμε το ταχύτερο με την νομοθετική μας βάση, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο. Αυτό που σα προτείνω, συνεπώ, είναι αύριο να ψηφίσουμε τις τροπολογίες και το ψήφισμα. Αντιθέτως να μην ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μόνο μία ψηφοφορία η οποία θα μείνει στην άκρη και γι' αυτό μπορούμε να ψηφίσουμε είτε τον Ιούλιο εφόσον έχουμε λάβει εντολή για να το πράξουμε και η παραδοσιακή γραμμή απασχόληση έχει ψηφιστεί ω οριζόντια γραμμή σε όλε τι επιτροπέ. Ή στο τέλο θα καταλήξουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση, όπου μετά από τον τριμερή διάλογο θα επανέλθουμε ενώπιον τη επιτροπή για να αναφέρουμε τα αποτελέσματα αυτού του τριμερού διαλόγου. Με λίγα λόγια, αυτό που σας προτείνω αύριο στην λίστα ψηφοφορίας ε, να ψηφίσουμε τις 120 συμβιβαστικές τροπολογίες μέχρι το γράμμα ταφ, ταφ, ταφ, ταφ, 4, 5 ταφ, αλλά να ψηφίσουμε στη συνέχεια για την πρόταση ψηφίσμα, νομοθετικού ψηφίσματος αλλά να μην ψηφίσουμε για το σύνολο της νομοθετικής πρότασης. Δηλαδή απλά η τελευταία ψηφοφορία δεν θα γίνει. Μέσα σε όλο αυτό το γραφειοκρατικό περίπλοκο χάος έχουν καταλάβει όλοι, γιατί μιλάμε και έχουν καταλάβει όλη τη θέση της Προεδρίας, όπως φαίνεται είναι. Καταπληκτικά λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Τρίτη παρατήρηση. Όπως γνωρίζετε, Όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Γιούτα Στάιντρο και είχαμε κινητοποιήσει τις νομικές μας υπηρεσίες επειδή ορισμένοι μας έλεγαν ότι κάνουμε πράγματα που δεν επιτρέπονται. Η νομική μας υπηρεσία μας έδωσε δίκιο. Έδωσε δίκιο στην πρόταση της συζητητριές μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με αυτή την άψη της νομικής υπηρεσίας αλλά ρωτήσαμε την νομική υπηρεσία και για μια άλλη διάσταση για ένα πράγμα που θέλει να πράξει και η ε, Κομισιόν όσον αφορά το Γιούρες. Η, η Επιτροπή μας όσον αφορά το Γιούρες. Στην περίπτωση του Γιούρες αρχικά πρόκειται για ένα κανονισμό για τον οποίο δεν είχε δικαίωμα απόφαση εξουσία απόφαση στο Κοινοβούλιο. Βάσει αυτού του κανονισμού λήφθηκαν ορισμένε πρωτοβουλίε για την υλοποίηση του προγράμματος Γιουρές. Σήμερα η Κομισιόν θέλει να αλλάξει αυτά τα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος Γιουρές χωρίς να επανέλθει στον ίδιο τον κανονισμό. Δηλαδή, ο ίδιος ο κανονισμός έχει αλλάξει νομική βάση. Δηλαδή, σήμερα εντάσσεται στη απόφαση. Θεωρούμε λοιπόν και μας ε, δίνει δίκιο η νομική υπηρεσία ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να αλλάζει τα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου εφόσον η νομική βάση έχει αλλάξει. Εάν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν θα αποταθώ στον Επιτροπό εξ ονοματός σας για να του πω ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να αλλάζει τα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος Γιούρες χωρίς ε, επίσημη τροποποίηση ή χωρίς ε, επαναφορά σε συναπόφαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του αρχικού κανονισμού που επιτρέπει τη λήψη αυτών των πρωτοβολιών. Σα ζητώ συγγνώμη που το κάνω αυτό στο όλο μελέτη τη Επιτροπής, αλλά καμιά φορά υπάρχουν έκτακτα περιστατικά που το επιτάσσουν. Ε, βλέπω ότι η κυρία Στάινρουκ φαίνεται να είναι ικανοποιημένη. Θα ψηφίσουμε έτσι λοιπόν αύριο για την εκθέση της κυρία Στάινρουκ για το σημείο 4. Δίνω το λόγο στην κυρία Μακιντάιρ. Όσον αφορά τις τροπολογίες για την εκθεσή της, για το σχέδιο γνωμοδότησής της, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και εμπορικές προοπτικές. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΤΡΕ. Κύριε Συγήτρια, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους σκιώδεις συζητητές για τη συνεργασία μας και για την υποστήριξή του που είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για όλους. Είμαι πολύ ικανοποιημένη για το ότι αναβάλαμε τις εξελίξεις για τον επόμενο μήνα. Καθέστε. Και πήγε το κείμενο για μετάφραση, επέστρεψε τέλη της προηγουμένης εβδομάδας. Και θεωρήσαμε ότι δεν γίνεται ανάλογα με τη σημασία του κειμένου να προχωρήσουμε όπως θέλουμε, οπότε ευχαριστώ όλους και ιδίως τον Φιλμπένιον από την περιφέρεια των Δυτικών Μίτλαντς και έχουμε εδώ 62 τροπολογίες. Και επίσης επεξεργαζόμαστε κάποιες συνδραστικέ τροπολογίες. Έτσι έχουν όλοι τον χρόνο να ασχοληθούν η μετάφραση ήταν πρόβλημα θέλω να σας πω ε, συγκεκριμένα τι έχουμε. Την ε, τροπολογία 23 του κυρίου Ποπάκη, το ελληνικό κείμενο, έτσι όπως μεταφράζεται και αποδίδεται στο ότι έτσι θα βελτιώσουμε την πρόσβαση των, ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και χρηματοδότησης. Θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να λέει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα είναι δυνατόν ε, και δεν το διορθώσαμε σε καμία φάση. Πρέπει να σου το πω αυτό, αν ε, τύχει να ρίξετε μία ματιά σε αυτές τις τροπολογίες. Άρα, ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά θα βοηθήσουν πάρα πολύ ε, οι τροπολογίες. Καλύτερα να τις στηρίξουμε όλοι και, και πάλι ευχαριστώ όλους. Ε, My colleague was uh, distracting me. Ο κύριος Μπένιον. Right, yes, I'd like to thank uh, uh, Mr. Συγγνώμη, μου είχε προσφέρει την προσοχή η συνάδελφος και να ευχαριστήσουμε την κυρία Μακιντάρ για την ε, εκθεσή τη. Όντως, η συνεργασία μα ήταν τέλεια για αυτή την έκθεση. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και την ε, πρόεδρο που συνεφώνησε να αναβληθεί η ψηφοφορία γιατί την Παρασκευή, αργά, ίσως, ίσως απόγευμα πέμπτης ελήφθησαν οι τροπολογίες, ε, την ώρα που επέστρεφα στην χώρα μου. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική έκθεση και άρα χρειάζεται χρόνος για να συζητηθεί όπως πρέπει. Έχουμε κάποιες τροπολογίες, έχουμε ε, πεδίο εφαρμογή κάποιων συμβαστικών τροπολογιών επίση. Έχουμε εδώ μια σειρά θετικών τροπολογιών. Πάντω, πρέπει να γίνουν συμβαστικές τροπολογίες, παράγραφος 2, 6, για τις 2 και 6. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Ε, είναι θετικό αυτό, γιατί έτσι συμβάλλουν περισσότερα σε αυτή την ε, έκθεση και όλα αυτά θα τα εντάξουμε σε κείμενο που θα μας βρει όλους σύμφωνος. Όντως, προκάλεσε προβληματισμό έτσι όπως μεταφράστηκε η τροπολογία από πάκι. Πάντως τώρα διορθώθηκε. Η τροπολογία ισότητα τώρα, ιδίως η 12 και 34 ε, θα μας απασχολήσουν. Στην 12 υποψιάζομαι ότι Τελικά θα συμφωνήσουμε με τις ουσίες, αλλά η αγγλική μετάφραση είναι δυσνόητη. Δεν προκύπτει με ακρίβεια αυτό που πρέπει. Άρα θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η γαλλική μετάφραση. Τώρα, πάλι της κυρίας Σουέτερ, η υπαριθμόν 34. Εδώ πρέπει κάτι να μας διευκρινίσει. Γιατί δεν ήξερε ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ υπάρχει. Υπάρχει. Ή το ζητάτε να συγκροτηθεί. Επίσης κάτι άλλο για τις 13 παραστημών 13 και 14. Για το κόστος χρηματοδότησης, πώς πρόσβαση χρηματοδότηση, ε, στο κείμενο εκδοχή του κειμένου κ. Μακητάρ τα έχει βάλει, δεν το περιλαμβάνεται εδώ, ε, ούτε, το, ούτε ζητάτε να απαλληφθεί, άρα είναι θέμα μήπως διατύπωσης. Καταρχήν συμφωνούμε στις 12.000, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει ε, κάτι, είναι να ανατεύσουμε αυτό που συμφωνήσαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Κοιτάξτε, καταρχήν, όλη, κάθε νομοθεσία μπορεί να είναι επαχθής. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ακόμα με το 18. Γιατί ακόμα και τα αναγκαία νομοθετήματα κάμια φορά είναι φραγμό σε μια δραστηριότητα. Εγώ εργαζόμαστε σε ΜΜΕ και, και ποτέ δεν ζητήσαμε να καταργηθεί κάποιο νόμο επειδή μα βαραίνει, επειδή μα εμποδίζει. Εντάξει. Κάμια μια φορά ε, κάποια πράγματα που βαραίνουν, που δυσκολεύουν, χρειάζονται. Καλύτερα μετά λέμε για ε, κάποια μέτρα που είναι χρονοβόρα, αλλά, φορούν τις καταστοιχές εργασίες και λοιπά, συμφωνούμε με αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, κύριε Ράινερ και τον κύριο Σίγκλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι όντως προσπάθησε στη συνεδρίαση να, <clears throat> με τους σκιώδεις να παρουσιάσει τα διάφορα θέματα ε, ιδίως ε, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο χαλαροί όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Βλέπουμε ότι εδώ ηγείται η Επιτροπή Ήτρε και το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει επιτρέπει αυτή τη χαλαρότητα, δηλαδή ε, τον χρόνο για να διερευνήσουμε ε, πιθανότητες ε, συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχουμε διάφορα θέματα. Καταρχήν την προστασία των εργαζομένων είναι πολύ βασικό να μην ε, ε, μπορέσουμε να ε, σκεφτούμε απλώς ότι θα χρειαστούμε μία, μία αγορά που να αποτελείται από τους εργαζομένους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να κοιτάζουμε πώς θα μειώσουμε την προστασία των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Επίσης, ε, όταν κοιτάζουμε να προσελκύσουμε εργαζομένους, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ε, γιατί δεν θα πρέπει να ε, πάμε χειρότερα αντί να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Στα πλαίσια αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, θα πρέπει ε, να προσέξουμε την ε, υγειονομική περίθαλψη αλλά και ολόκληρη την άποψη της κοινωνικής απασχόλησης και επίσης ένα άλλο θέμα που θέλω να τονίσω είναι η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν πρέπει να είναι κανείς καινοτόμος για το μέλλον και ε, η διτή εκπαίδευση κατά τρόπον ώστε οι νέοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση για μετεκπαίδευση ε, και στάζ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς αυτή η δυνατότητα να περιορίζεται από περιοριστικούς οικονομικούς παράγοντες. Ακριβώς οι νέοι πρέπει πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εργασία πιο εύκολη και υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ καινοτόμες και μπορούν ε, να δρομολογήσουν ε, βασικά οικονομικά θέματα και ε, εκεί η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει επίσης να περιληφθεί στη γνωμοδότηση την οποία διατυπώνουμε. Ευχαριστώ η κυρία Σανκλέρ και η κυρία Σρέντερ και έτσι κλείνουμε τη λίστα των ομιλητών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Μακεντάερ για αυτή τη γνωμοδότηση. Δεν θα, θα σας κάνει έκπληξη. Δεν ε, έχω αντίρρηση με τα περισσότερα από όσα λέει. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια το να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομέσες επιχειρήσει όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είμαστε και οι δύο από το West Midlands, ε, ε, έχουμε τον ίδιο αριθμό ψηφοφόρων και εγώ του συναντάω σε εβδομαδιαία βάση και όπως και ο κ. Μπένιαν, θα ήθελα να καταλα... είναι πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο στο West Midlands, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα σας έρχεται εδώ, κυρία Μακιντάερ λέγοντας ότι μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και εδώ ε, δίνεται μια γνωμοδότηση. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι το συντηρητικό κόμμα δεν έχει αρκετά μέλη σε αυτήν την επιτροπή. Αυτό είναι, είναι πολλά λόγια αυτά που λέτε, αλλά έλλειψη δράσης. Και οι δυο μα το 2009 ε, παραστήκαμε στην Ευρωπαϊκή Εκλογή, στη συνεδρίαση εκλογής της, ε, ε, του συνασπισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και θα θυμάστε ότι τα μανιφέστο που μας έδωσαν όλοι Αριθμό 1, σας παρακαλούμε, όχι άλλη παρεμβολή η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μετά από τρία χρόνια, όλο και περισσότερη νομοθεσία ευρωπαϊκή επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ο κ. Όσμπορν είχε μιλήσει για τις επιπτώσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν μίλησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το πραγματικό πρόβλημα. Μίλησε για το τι θα κάνει η δική του κυβέρνηση αλλά δεν μίλησε για τα μέρη, για τους τομείς στους οποίους δεν έχει εξουσία και εσείς όπως ο κ. Μπέριν ε, ως εκπρόσωποι του κυβερνητικού κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου θα έπρεπε να, ε, να, να πείτε την άποψη διότι αποτυγχάνετε. Δίνω το λόγο στην κυρία Σρέντερ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην κυρία Σενκλέρ ότι οι αναπληρωτές αυτής της Επιτροπής αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι και δεν υπάρχει διακρίση μεταξύ ε, μελών και αναπληρωτών. Εφαρμόζουμε μη διακριτική μεταχείριση και σε αυτόν τον τομέα. Θα δώσω δύο παραδείγματα για το κόμμα του ΕΕΛΚ. Ο κ. Σογκόρ είναι εισηγητής για ένα πολύ σημαντικό φάκελο σε θέματα στατιστικά και η κυρία Σιπέλ ε, των Σοσιαλιστών είναι εισηγήτρια για ένα εξίσου σημαντικό φάκελο την πρόσβαση στις δημοσίες συμβάσεις. Προτείνω λοιπόν να σταματήσουν αυτού του είδους οι παρατηρήσεις που δεν έχουν θέση σε αυτή την Επιτροπή. Δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση, κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την εργασία που έκανε. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση χωρίς να υπάρχουν τροπολογίες στη διάθεσή της διότι εγώ τις τροπολογίες μου τις έχω διατυπώσει στην μητρική μου γλώσσα τα γερμανικά γι' αυτό και ενδέχεται να έχουμε προβλήματα μεταφράσεως. Εγώ δεν ε, έχω ακόμη ελέγξει αν το κείμενο με νόμο έχει ε, μεταφραστεί σωστά προς τα αγγλικά για να απαντήσω στις ερωτήσεις της συναδέλφους. Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι λογικές και ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα επικοδομητικό αποτέλεσμα. Ε, Βεβαίω, ε, φαντάζομαι αλλά το θέμα είναι ότι εάν είμαστε όλοι ίσοι, τότε γιατί έχουμε διαφορετικό χρώμα κάρτας. Τι είναι η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Όχι, λέει η κυρία Μπερές, μόνο την ότι ψηφοφορία υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά στην μεταχείριση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιτροπή. Μπορείτε να λάβετε εκθέσεις, μπορείτε να μιλάτε, μπορείτε όλα τα σας ενημερώνω με μεγάλη μου ικανοποίηση επ' αυτού. Κύριε Μακιντάρη, τώρα ερωτήσαμε την εκθεσή της. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι έγινε αυτή η αναβολή της ψηφοφορίας για το σύνολο της έκθεσης, διότι η Ήτρα ε, και εκείνη ανέβαλε την ψηφοφορία. Και η μετάφραση των τροπολογιών, όπως είπε ο κύριος Έγινε έτσι γιατί ήταν τέτοιε οι συνθήκε εργασία μα, μια που στην τελευταία ολομέλεια είχαμε πολύ μικρό διάλειμμα μέχρι την επομένη ολομέλεια και έτσι δεν μπορέσαμε να κάνουμε όπω πρέπει τη μετάφραση. Οπότε λόγω αυτή τη κατάσταση έγινε η ενοβολή και έτσι ξεπεράσαμε τι δυσκολίε Θα δευτερολογήσω τώρα κυρία Συγήτρια για να ολοκληρωθεί το θέμα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για να επανέλθω σε δύο πράγματα και που υπόθηκαν. Η κυρία Σινκλέρ θα ενδιαφέρεται να μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ε, υποστηρίζει την παρούσα γνωμοδότηση. Έχω ένα δελτίο τύπου τους ε, σχετικά με αυτό. Συνεπώς μην θεωρείτε ότι δεν έχουμε λάβει την υποστήριξή τους. Και ε, εκπροσωπούν ε, τις διάφορες ομοσπονδίε, όπως και την FSB, η οποία είναι αυτή στην οποία εσεί αναφερθήκατε. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να περικόψουμε την προστασία των εργαζομένων και να έχουμε δύο κατηγορίες εργαζομένων. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα όπου η μείωση της γραφειοκρατίας έκανε μια μεγάλη διαφορά. όσοι ε, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ένα περίπλοκο σύστημα για την πληρωμή ατόμων όπου έπρεπε να συμπληρώσουμε έντυπα, να αφαιρέσουμε το φόρο και την ε, εθνική ασφάλιση, ε, την κρατική ασφάλιση και δαπανούσε κανείς πολύ χρόνο για όλα αυτά. Η κυβέρνηση μετά εξέδωσε ένα CD που το βάζει στο κομπιούτερ και κάνει όλη τη δουλειά. Συνεπώς ε, δουλειές που ε, μου έπαιρναν μισή μέρα τώρα μου παίρνουν μισή ώρα. Αυτού του είδους τα πράγματα θα πρέπει να επιτυγχάνουμε σε όλη την Ευρώπη. Διότι αυτά διευκολύνουν την καθημερινή μας ζωή και ε, βοηθούν στην πρόσληψη ανθρώπων από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία θα ήθελα να επιδιώξω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ του ε, σκιώδεις ηγητέ για τη συνεργασία τους και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε, ικανοποιητικού για όλου σε ικανοποιητικούς Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε την εκθέση, την γνωμοδότησή σας στις 10 Ιουλίου. Περνώντα στο σημείο 5 τη ημερησία διάταξη θα πρέπει να δούμε τη διάρθρωση μεταξύ αυτών των δύο σημείων, τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο σημείων, διότι η γνωμοδότηση τη οποία είστε συντάκτρια είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε και φτάνοντα στο σημείο 5, όπου εγώ είμαι η συγκήτρια, εκ μέρους όλων σας ε, όσον αφορά το ψήφισμα για τις συνέπειες για την απασχόληση της ελασχιστοποίησης του κανονιστικού φόρτου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. το σκεπτικό των συντονιστών για αυτή την πρωτοβουλία ως προφορική ερώτηση και ως ψήφισμα ήταν ε, να απαντήσουν στην ανακοίνωση της Κομισιόν όχι μόνο από απόψη όσον αφορά τις ανησυχίες της ΣΥΤΡΕ αλλά και για να δημιουργηθεί μια βάση ώστε να αναφέρουμε τα ζητήματα υγείας και ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και στις δομές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε μία κοινή προσέγγιση, επειδή θα ήταν παράδοξο αυτή η Επιτροπή να ψηφίσει την έκθεση McIntyre και το ψήφισμα και το προφορικό ερώτημα. Θα πρέπει να τα λάβουμε λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία ως ε, ενιαία Υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποιες τροπολογίες για την προφορική ερώτηση που δεν θέτουν κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά το ψήφισμα, υπάρχουν, έχουν υποβληθεί 49 τροπολογίες. Θα επικοινωνήσω φυσικά με τους συντακτές των τροπολογιών για να καταφέρουμε να βρούμε συμβιβασμούς και ειδικότερα τον συντονιστή διότι αυτός θα πρέπει να συντονιστεί για να συντονιστούν οι σκιώδεις συζήτητες, αλλά ήθελα να αναφέρω κάποιες τροπολογίες για τις οποίες θεωρώ ότι έχουμε κάποιες ε, διευκρινήσεις που απομένουν να γίνουν. Βλέποντας τις τροπολογίες 17 και 18, 17 της κυρίας Μακιντέρ και 18 του κυρίου Κρίστενσεν και Λούδβιξον, που αφορούν τις συνθήκες προστασίας των εργαζομένων βλέπω ότι έχουμε δύο δικροόμενες προσεγγίσεις. Θα χρειαστεί λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία η οποία θα μας επιτρέψει να ορίσουμε τη θέση της Επιτροπής. Δεν θα σας κάνει έκπληξη το να σας πω ότι κατά την απόψή μου η τροπολογία 18 είναι αυτή προς την οποία θα πρέπει να προσανατολιστούμε θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία δεν πρέπει να θεωρείται διοικητικός φόρτος ε, που δεν μπορούν να ε, υποστηρίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετέχουν τις τροπολογίες 36, 37, 38 και 39 που αφορούν ε, την παροχή κινήτρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να οργανώνονται για προσαρμοσμένη αντιπροσώπευση, κροσόπηση των εργαζομένων και την δημιουργία δομών που επιτρέπουν ε, τη λειτουργία ενός κοινωνικού διαλόγου και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τέσσερις τροπολογίες από την κυρία Μακιντήρ, τον κύριο Ρή, τον κύριο Μπενίον από τους φιλελεύθερους και την κυρία Σρέντερ για τους πράσινους. Ε, διακρίνω στοιχεία στα οποία, βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, αλλά θα χρειαστεί συναπόφαση μεταξύ μας. Θεωρώ ότι το ενδιαφέρον που έχει ένα τέτοιο ψήφισμα για την Επιτροπή μας είναι να προχωρήσουμε κάποια πιόνια. Εάν μείνουμε στο να μην αλλάξουμε τίποτα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν προχωρήσουν σε κοινωνικό διάλογο, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η παράγραφος 11 ουσιαστικά προωθεί την ιδέα ότι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούμε να έχουμε αμοιβαίο κοινωνικό διάλογο που θα επιτρέψει την εξέλιξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και την προσαρμογή του σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στη συνέχεια όσον αφορά την παραγραφό 9 Υπάρχει το ζήτημα της κοινωνικής ε, προστασίας και να δούμε ποιες συνθήκες επιβάλλει αυτή η νομοθεσία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί θα χρειαστούμε διαιτησίες ε, διότι υπάρχουν τροπολογίες Εκεί θα χρειαστεί μια συζήτηση εντό των σοσιαλιστών, διότι έχουμε τροπολογίες Ρέγνερ και Στάινρουκ και από τον κύριο Κρίστενσεν και από τον κύριο Λούντβιξον. Θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για, μεταξύ αυτών των δύο τροπολογιών. Τώρα, μετά την παράγραφο 9, η τροπολογία 61 της κυρίας Ήρς, που επιμένει στην αναγκαιότητα Άρση των διοικητικών εμποδίων, των διοικητικών φραγμών, κυρίως όσον αφορά την πρόσληψη εργαζομένων από τρίτες χώρες το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις δικές μας ανησυχίες ε, σε αυτή την Επιτροπή σε όλες τις ομάδες για την ισο... ότι η ίση εργασία πρέπει να αντιστοιχεί σε ίσα δικαιώματα. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελα να σας αναφέρω όσον αφορά αυτές τις 49 τροπολογίες. Ο κύριος Μπένιον μου έχει ζητήσει το λόγο, τον οποίο το δίνω πολύ ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Όπως είπατε, αυτό το θέμα σχετίζεται με το μέρος προηγούμενο. Κατά τη γνώμη μας, και η προφορική ερώτηση αλλά και το ψήφισμα είναι αξιόλογο. Και θα τα βελτιώσουμε με τις τροπολογίες για απλούστευση κανόνων, μείωση γραφειοκρατίας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξορισμού επιβλαβή. Δηλαδή. Άρα θα πρέπει κάπως να χτενίσουμε αυτές τις ε, αρνητικές διατυπώσεις και όπως και πριν, είπαμε θα πρέπει να έχουμε η νομοθεσία, απλή και αποτελεσματική. Αν κάτι είναι υπερβολικά περίπλοκο και εμποδίζει, τότε είναι φραγμός στις ΜΜΕ. Γιατί οι, η manager στις ΜΜΕ πασχίζουν εύκολα να μάθουν τους νόμους που διέπουν την ΜΜΕ. Άρα θα πρέπει να γίνει απλή νομοθεσία, εύκολο να εφαρμοστεί και έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε αυτά που σκοπεύουμε, δηλαδή ασφάλεια και κατοχήρωση των γενικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα πούμε και με θετικό τρόπο και άλλες τροπολογίες. Επ' αυτού ελπίζω θα βρούμε τη μέση οδό, συμβαστική τροπολογία, γύρω στο 10, που λέει για απλούστευση σε επίπεδο των μελών. Επίση, πάρα πολύ θετικά βλέπω το 11, που λέει την εκπροσώπηση των ΜΜΕ στον γενικό διάλογο. Και έχουν πάρα πολλέ τροπολογίε, αλλά νομίζω ότι θα είναι η κατάληξη πάρα πολύ θετική. Γενικά, θετικά βλέπουμε ότι λέει για την εκπροσώπηση ε, των τον ΜΜΕ, τον Γενικό Διάλογο. Υπάρχουν κάποιοι φορεί που τις εκπροσωπούν, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δεν υπάρχουν να φτιάξουμε και που λέμε για την ε, Ομοσπονδία των ΜΜΕ. Υπάρχει τέτοια οργάνωση, αλλά έχουμε και την CBI για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά εκεί ανοίγουν και κάποιες ΜΜΕ. Επίσης, έχουμε πολλούς, πολλούς εμπορικούς φορείς και για τους γεωργούς ακόμη, η οποία είναι παρελθόντως πολύ αποτελεσματική και δραστήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε καινούργιε μορφέ εκπροσώπηση, αλλά θα πρέπει στο κοινό διάλογο να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσε. Όπως είπε και η Πρόεδρος. Θεωρώ ότι είναι θετικό να υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να ακούγονται οι απόψεις όλων τους κοινωνικούς εταίρους γιατί προσφυστηρούμε ότι οι μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν και ότι έχουν περιθωριοποιηθεί οι ΜΜΕ. Άρα θα πρόκειται για θετική αλλαγή. Αν γίνουν όλα αυτά τα οποία προτείνει η έκθεση. Και νομίζω ότι η Γενική Συνένεση συγκεντρώνεται γύρω από αυτό το κομμάτι του κειμένου. Πρόεδρος, αν δεν υπάρχουν άλλοι ε, ομιλητές, να το τελειώσουμε με αυτό το θέμα και όπως είπαμε και προηγουμένω στην εισαγωγή. Η κυρία και οι θα γίνει μια συζήτηση, ούτως ώστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των δύο κειμένων και θα γίνει κάποια στιγμή η ψηφορία. Στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. Τώρα πάμε στο σημείο υπαριθμών 6 και τον λόγο έχει τώρα η κυρία Ιώτοβα. Αφορά την εξέταση των τροπολογιών για την έκθεσή της. Επιτροπή Γυναικών. Όσον αφορά τι θέσει των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών. Έχει το λόγο κυρία Ισηγήτρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω τώρα στα βουλγάρικα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες που είχαν λίγο χρόνο για να προετοιμαστούν για αυτήν την ε, ε, γνωμοδότηση είχαμε 38 τροπολογίες και μπορέσαμε την περασμένη εβδομάδα να καταλήξουμε σε ορισμένες συμβιβαστικές 19 ε, τον αριθμό και οι υπόλοιπες τροπολογίες δεν μας προβληματίζουν εκτός από δύο με τις οποίες δεν συμφωνούμε ε, το, την τροπολογία 6 και 34. Στην τροπολογία 6 αναφερόμαστε στις πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας οι οποίες απορρίπτονται και ε, ε, θεωρούν ότι διαταράσσουν την ε, συμβατότητα εργασίας ε, και οικογενειακής ζωής. Γι' αυτό και λέει το αρχικό κείμενο ότι οι εργαζόμενοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευέλικτες μορφές ε, εργασίας θα έπρεπε να τις προτιμήσουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ευέλικτο χρονικό πλαίσιο εργασίας και άρα θα μπορέσουν να απασχοληθούν περισσότεροι ελεύθεροι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή ενώ όταν υπάρχουν ε, συνηθισμένες συλλογικές συμβάσεις ε, από που εφαρμόζονται ε, υπάρχει και η πλήρης ε, υγειονομική και κοινωνική κάλυψη και αυτή θα έπρεπε να ισχύσει και εδώ. Στην ε, άλλη τροπολογία αναφερόμαστε εις γυναίκες που έχουν παιδιά τουλάχιστον 12 ετών πράγμα το οποίο αντιφάσκει με τη βασική σκέψη και μπορεί να αποτρέψει τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να εργαστούν. Λέγεται δε ότι ε, τα μέτρα εξοικονόμησης ε, θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερο τις γυναίκες που εργάζονται στα κράτη-μέλη. Οι γυναίκες πάντοτε είναι σε δυσμενέστερη θέση και χρησιμοποιούνται σε πιο προσωρινές θέσεις εργασίας χωρίς να μπορούν να χαίρουν τις ίσεις αμοιβή για την ίση εργασία. Επίσης ε, ε, επηρεάζονται και απειλούνται από περικοπές στις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και εμείς θα θέλαμε να διατηρηθεί το αρχικό κείμενο το οποίο λέγει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να ε, να απελούνται σε περίπτωση ε, περικοπών εργασίας. Το 2007 στην έκθεση, στην, ε, για την έκθεση η οποία είχε καταρτιστεί ε, είχε γίνει μία μελέτη για την ισότητα αντιμετωπίσεως στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών και είχε, είχε εξετάσει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων εκ των οποίων 17% είχαν πει ότι ε, είχαν ε, ε, απασχοληθεί στον τομέα των υπηρεσιών πράγμα το οποίο σημαίνει 3,5 εκατομμύρια άτομα τα οποία ουσιαστικά εργαζόντουσαν σε οικιακές εργασίες χωρίς να είναι δηλωμένες όπως παραδείγματο χάρη στο Βέλγιο όπου δεν υπήρχε, ε, υπήρχε ε, κοινωνική κάλυψη. Στο Βέλγιο παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα καλό σύστημα όπου το ίμιση των, της κοινωνικής ασφάλειας καλύπτεται από το εργοδότη και το άλλο ήμιση από το κράτος. Είναι ένα καλό παράδειγμα. Σας ευχαριστώ για τι ορπολογίε σας και παρακαλώ να σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ε, ότι το μήνυμά μας σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε κάποια σημεία. Δηλαδή Στη παράνομη εργασία, στη συνέχεια στην υποστήριξη των επιχειρήσεων, στις ε, οικιακές βοηθούς, στις γυναίκες που εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και θα πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτό το σύστημα του burnout το μήνυμά μας, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτά τα σημεία. Φυσικά υπάρχουν τροπολογίες που δεν υποστηρίζονται από όλους. Αλλά πιστεύω ότι όταν έχουμε αμφιβολίες ε, θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ε, βάσει της τροπολογίας 6 συμφωνώ και συμφωνούμε με το συμβιβασμό. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κ. Πουπάκης είναι εδώ θα ήθελα να μας πει τι θεωρεί ότι βρίσκεται πίσω από την τροπολογία 18 διότι διάβασα πολλά αλλά αυτό το μοντέλο για το οποίο μιλάει τι, τι, μοντέλο, τι υπάρχει πίσω από αυτό της ε, της εργασίας αυτό ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Και συμφωνούμε με το συμβασμό φυσικά. Η 18 δεν είναι ποτέ. Qu'est-ce qui parle Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Γενικά, είναι ικανοποιητική αυτή η Έχετε συμφωνήσει με τις τροπολογίε και συμφωνούμε με το ότι η κυρία ε, είπε και η κυρία Ιώτοβα ε, να φέρει πίνη ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες ρυθμίσεις εργασιακέ ευέλικτε και ότι αυτό από μια μεριά μπορεί να αποτελέσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν έχουμε συνέχεια αλλαγέ, έχουμε δύσκολε ώρε και δεν μπορεί κανεί να έχει λέγει όσον αφορά τι βάρκε που θα κάνει και δεν μπορεί τέλο πάντων το επαγγελματικό βίο να τον ρυθμίσει. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί η άλλη νομίσματο να είναι το θετικό γιατί έτσι κάποιο μπορεί να δουλέψει έτσι περισσότερο όταν βολεύει, να δουλέψει λιγότερο όταν δεν βολεύει. Ε, Α πούμε για του διαζευμένου γονεί που του βολεύουν οι, οι, οι περίεργε ώρε εργασία όταν τα παιδιά είναι με τον άλλο πρώην Οπότε θα πρέπει τελικά να έχει την επιλογή ο εργαζόμενο και θα πρέπει να ασκεί έλεγχο όσον αφορά τι ρυθμίσεις της ε, εργασίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ευελιξία, είναι κάτι το θετικό. Επίσης έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες τη ΓΚΟΕ με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Ας πούμε η υποχρεωτική εξαίρεση για του εργαζόμενου τη νύχτα Ε, αυτό δεν είναι. Κάποιοι το θέλουν γιατί θέλουν να συνδυάσουν κάποια άλλα πράγματα. Άλλε υποχρεώσει, επίση οι ελάχιστε προδιαγραφέ, ε, να καταπολεμήσουμε την παρανομή εργασία, την τη εργασία. Τα ελάχιστα, ελάχιστε ρυθμίσει για τι υπηρεσίε. Ούτω ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά του οι εκεί εργαζόμενοι στι υπηρεσίε. Να προστατεύσουμε του πιο ευάλωτου επομένω. Εκεί τα καταψηφίζουμε κάποιε από τι τροπολογίε, αλλά είμαστε υπέρ των περισσότερων. Θεωρούμε πάρα πολύ ικανοποιητικό το έργο τη κυρία Διώτοβα. Κύριε Ποπάκη, θέλετε το λόγο. Όχι απλά επειδή αναφέρθηκε το όνομα μου και στη συγκεκριμένη τροπολογία που καταθέσαμε, Εμεί απλά θέλαμε να τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η διαφύλαξη δηλαδή, η ενίσχυση τη υγεία στην ασφάλεια και εργασία. Και έχουμε συμφωνήσει με τον συμβασμό. Ε, Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα ρουμάνικα με την αδειά σας. Ε, η έκθεση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εξετάζει έναν τομέα όπου οι γυναίκε αποτελούν την πλειοψηφία. Ταυτόχρονα πρόκειται για έναν τομέα που παρέχει δουλειά σε γυναίκες παρότι έχουν περάσει 150 χρόνια από τη βιομηχανική επανάσταση φαίνεται ότι οι γυναίκες ακόμη και σήμερα καταλήγουν με αυτού του είδους τις εργασίες και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συμφιλειώσουν τις ε, ε, επαγγελματικές και οικογενειακές ζωές τους όπως υπογραμμίζει η συγγήτρια υπάρχει δυνατότητα ευέλιξης λύσης και προσέγγισης ώστε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν τις, τα καθήκοντά τους ε, στον επαγγελματικό και στον οικογενειακό τομέα. Ε, ταυτόχρονα χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι στις συμβιβαστικές τροπολογίες η ιδέα ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμφιλειώσουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές ζωές τους διατηρείται. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για αυτό και τη θεωρώ πολύ θετική ένδειξη και χαίρομαι επίση που μία από τις δικές μου ιδέες που υπέβαλα με τροποποίηση όσον αφορά τους πιο ευάλωτους ανθρώπους έχει επίσης διατηρηθεί. Η συγγετρία και οι υπόλοιποι ενδιαφέρομενοι θεώρησαν ότι ήταν ωφέλιμη αυτή η συμβολή. Θεωρώ ότι αυτή η εκθέση είναι πολύ σημαντική. Υποστηρίζω τι τροπολογίε, ε, όπω απορρέουν από τη διαπραγμάτευση και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Έχουμε ολοκληρώσει τη λίστα των ομιλητών και δίνω το λόγο στην εισηγητριά μας. Δεν χρειάζεται, όχι. Ωραία λοιπόν, υπό το πνεύμα αυτό μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο για τη γνωμοδότηση της κυρίας Ιώτοβα ώστε να λυθεί η ψηφοφορία μας αυτή ε, υπόψη στην Επιτροπή ΦΑΜ για την ψηφοφορία του στις 10 Ιουλίου. Περνάμε στην έκθεση του συναδέλφου Όλε Λούντβιξον για την εξέταση των 60 τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδότησης που συντάσσουμε για το πρόγραμμα εκπαίδευση, κατάρτιση και Ευρώπη 2020. Κύριε Ισήτη, έχετε το λόγο. Ευχα... Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες είναι επικοδομητικές και επικοινωνούνται προ τη σωστή παρόμοια κατεύθυνση. Έχουμε λάβει 60 τροπολογίες σύμφωνα με τι περισσότερε από αυτέ. Στο απόγευμα στείλαμε 10 προτάσεις βεβασμού στου κοιόδη εισηγητές και στην γραμματεία των, στις γραμματείες των ομάδων και αναμένουμε απαντήσεις. Το σχέδιο καλύπτει 39 τροπολογίες και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που καλύπτονται με άλλες μορφές διατύπωσης, σε άλλες ε, τροπολογίες. Αλλά ήταν δύσκολο το να καταλήξουμε έγκαιρα σε αυτούς τους συμβιβασμούς. Ε, την αγγλική μετάφραση τη λάβαμε μόλις τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας και μετά χθε. Ε, όλες οι μεταφρα... τα κείμενα μεταφράσεις, στάλησαν μεταφράσεις συγγνώμη του κειμένου, νομίζω, εκτός από τα δανέζικα. Είναι δύσκολο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας εδώ όταν έχουμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχω λοιπόν μια πρόταση να κάνω, ίσως να αναβάλουμε λίγο την ψηφοφορία μέχρι την συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου στο Στρασβούργο ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε σωστά σε αυτό. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σωστά με τους κοιόδης συζητητές, να συζητήσουμε γενικά και μερικοί από τους συζητητές δεν έχουν καταφέρει να διαβάσουν ακόμα σωστά το κείμενο και να μελετήσουν σωστά τις τροπολογίες. Όσον αφορά τους συμβιβασμούς που έχουν ήδη ε, διατυπωθεί, πρέπει να πω Ο Πρώτος συμβιβασμός αφορά την προνομιακή μεταχείριση της εκπαίδευσης ε, όσον αφορά την κρίση ως επένδυση για το μέλλον. Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδης δικαίωμα. Αυτό καλύπτει τις τροπολογίες 1 έως 34. Όσον αφορά το συμβιβασμό 2, μιλάμε για επένδυση σε ποιοτική εκπαίδευση. Αυτή μπορεί να συμβάλλει στο να μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Επίσης βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτούν τα σωστά προσόντα για πολλές διαφορετικές εργασίες. Με αποτέλεσμα περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης όσον αφορά το, 2 και μιλάμε, το σημείο 2 και μιλάμε για τις ε, τροπολογίες 6, 7, 8 και 9. Αυτή είναι ο συμβιβασμός 2. Ο συμβιβασμός 3 αφορά την προσαρμογή των πρακτικών στην αγορά εργασία. Χρειαζόμαστε περισσότερε συνδέσει μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και εταιριών. Πρέπει να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία. Θα μα βοηθήσει στο μέλλον. Ο συμβιβασμό επίση 3 αφορά τις τροπολογίες 10, 11, 14, 18, 19, 37 και 48. Συμβιβασμός 4. Τώρα οι προκλήσει εδώ αφορούν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε για το μέλλον και πώς ε, συντεριάζουμε την εκπαίδευση με τις μελλοντικές ανάγκες απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι που προκύπτει συχνά στην αγορά εργασίας, διότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι άνθρωποι δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτός ο συμβασμός καλύπτει τροπολογίες 15, 21, 22, 23, 24 και 25. Ο συμβιβασμό 5 εδώ αφορά τη σπουδαιότητα των επαγγελματικών καταρτήσεων για νέους και ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να καταλήξει σε ελάχιστα πρότυπα για αυτόν τον τομέα. Καλύπτει τις τροπολογίες 29, 31, 32, 33 και 36. Τροπολογία 6 είναι πολύ σημαντική για το μέλλον. Η διαβίου εκμάθησε. Όσοι σήμερα εργάζονται ήδη πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν να μαθαίνουν στη δουλειά τους. Εγώ ως διαπραγματευτής έχω συμμετέχει εκ μέρους διαφόρων ανθρώπων που έχουν χάσει τις δουλειές τους λόγω υπερβάλλοντος προσωπικό όταν δούλευα στη Βόλβο και το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας αφορούσε ανθρώπους που πάντα έκαναν την ίδια δουλειά. Ανέκαθεν και ποτέ δεν έλαβαν επιπλέον κατάρτιση ούτε σε τεχνολογικά ζητήματα. Είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση και καλύπτει αυτός ο συμβασμός αυτή η συμβαστική της τροπολογίας 41, 42, 43 η συμβιβαστική 7 αφορά ανθρώπου που εγκαταλείπουν το σχολείο και τη δημιουργία μια αρχική σύνδεση μεταξύ των αρχικών και των πιο προηγμένων σταδίων εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνέχεια. Όταν τα παιδιά, οι μαθητέ εγκαταλείπουν το σχολείο υπερβολικά νωρί, δεν αποκτούν τι κατάλληλε ικανότητε και έτσι δεν είναι ελκυστική για την αγορά εργασία, για του ε, εργοδότε. Αυτό είναι φυσικά μια πολύ σημαντική πτυχή. Αυτή η συμβιβαστική καλύπτει την τροπολογία 38 και εκεί έχω προσθέσει και κάποιο κείμενο ο η συμβιβαστική 8 αφορά τη σπουδαιότητα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Το σκεπτικό είναι να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι από πρώιμο στάδιο ώστε να μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα καλύπτει τις τροπολογίες 45, 55 και 60 η συμβιβαστική 9 αφορά τη σπουδαιότητα δημιουργία συστημάτων επαγγελματικών προσόντων για άτυπη και επίσημη εκπαίδευση. Εδώ μιλάμε για τις τροπολογίες 16, 50 και 51. Για τη συμβιβαστική 8 μιλάμε για την εξωτερική διάσταση που χρειάζεται ενίσχυση. Έχουμε λοιπόν αυτούς τις συμβιβαστικές που ουσιαστικά καλύπτουν τις περισσότερες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. παρότι δεν ανέφερα όλες τις τροπολογίες, έχουμε αλλάξει ε, τη διατύπωση ορισμένων συμβιβαστικών ώστε να τις καλύψουμε. Ε, έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να καταλήξουμε σε συμφωνίες όσον αφορά τις συμβιβαστικές και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό αυτό Είμαι ευγνώμων σε ό, για όλους τους κοιόδους εισηγητές για τη συμμετοχή τους, για τα σχόλιά τους, τις απόψεις τους. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να διαβάσω τις συμβαστικές τροπολογίες, αν χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Εάν αυτό συμβαίνει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω email και να μείνουμε σε επαφή με αυτόν τον τρόπο, εάν το επιθυμείτε. Για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω το εξή. Για να κάνουμε σωστή δουλειά σε αυτή την επιτροπή πρέπει να φροντίσουμε όλοι να έχουν στη διάθεση του τα εργαλεία. Ο εισηγητή χρειάζεται τα εργαλεία, αλλά το ίδιο και οι σκιώδει εισηγητέ. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να μιλήσουμε με τις ομάδες μας, διότι ο χρόνος που έχουμε εδώ απλά δεν αρκεί. Προτείνω λοιπόν να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την 5η Ιουλίου, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε σωστά για αυτό το εξάλλου πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, προτείνεται αναβολή της ψηφοφορίας για τις 25, τις 27 ή τις 5 Πεντηριλίου. Για τις 5 Ιουλίου. Για τις 5 Ιουλίου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ αυτή δεν τα είπα τόσο σαφώς. Καλά λέει πρόεδρος. Ε, στις 27, έτσι καλώς δεν είχαμε συνάντηση αυτό και τα Ο Κύριος Σόγκορ και κατόπιν ο κύριος Μπένιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε, Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έχουμε εδώ ένα σχέδιο εκθέσεως ιδέας πρωτοβουλίας. Πρόκειται για σημαντικό πρόγραμμα. Πρόκειται για τις εγγύσεις που θα κατοχυρώσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόκειται για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό είναι η Ευρώπη του μέλλοντο. Και εγώ ε, έχω υποβάλει κάποιε τροπολογίε. Γιατί βέβαια από την άλλη μεριά είχαμε πρόβλημα το ότι άργησαν πάρα πολύ να έρθουν ε, οι διαφορετικέ γλωσσικέ ειδοχέ στο κείμενο. Πάντω βλέπετε από τι τροπολογίε ότι όλοι είμαστε καλόπιστοι, όλοι πιστεύουμε θα τα βρούμε και <clears throat> ότι τελικά Νομίζω ότι με το σωστό ρυθμό κινηθήκαμε παρά ε, τη βιασύνη που μας οδήγησε, που οδήγησε τον κύριο Σιγητή να ζητήσει αυτήν την αναβολή. Δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε ε, πάρα πολύ. Βλέπουμε στο γόνατο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπένιον, λέει πρόεδρος. Απλώς να σας πω ε, εδώ για την κυρία Μάνων. δεν πρέπει να πάει κάπου Λέει λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι τον εισηγητή. Ε, και εγώ θα ήθελα, μας λέει, να σας πω κάτι για τις συμβασικές τροπολογίες. Συμφωνώ με τις υπαριθμών 1, 3 και 6. Ή στην υπαριθμών 2, η συνάδελφος θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μιλήσουμε για υψηλότερη ποιότητα, όχι για καλύτερη ποιότητα και μετά στο τέλος λέει να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος έχει τις δεξιότητες για καλύτερες ε, δουλειές ε, και έτσι να έχουν ασφάλεια στην απασχόληση, οπότε καλύτερα να πούμε ε, ποιότητα και βιώσιμη φόρο απασχόληση, γιατί είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε άλλα νομοθετήματα στη συμβαστική υπάρχει τέσσερα λέει, στην φράση που αναφέρει βασική και το βασικό πρόβλημα ε, της δομικής διαρθρωτική ενεργείας είναι ότι δεν ταυτίζεται η κατάρτιση με τι δουλειέ. Ε, λέει ότι θα πρέπει ε, να δούμε πώς τον επαγγελματικό προσανατολισμό που είναι πιο σημαντικό από την επαγγελματική κατάρτιση ε, θεωρεί είπαμε, ότι αυτό λείπει από την πρόταση. Η τελευταία φράση δε λέει ότι χρειάζεται ε, καταρτισμένους, με ειδικέ δεξιότητες εργαζομένους, θέλουν να στηριχθούν οι τέχνες οι παραδοσιακές. Ε, λέει ότι εδώ πέρα πρέπει να επαναδιατυπωθεί γιατί πλεονάζει το κείμενο και στο 7 λέει ότι είναι κάπως ασαφής διατύπωση και θα πρέπει επίσης να τη χτενίσουμε. Ε, Ευχαριστώ. Δεν έχουν εγγραφεί άλλοι ομιλητέ. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας αν και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ανάγκη σε αυτή τη φάση. Παρουσιάσατε τις συμβαστικές τροπολογίες, δεν έχουν λάβει ακόμα πλήρη γνώση όλοι οι συνάδελφοι. Ε, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ώστε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την 5η Ιουλίου. Θα είναι τρομακτική εκείνη σε ψηφοφορίε εκείνη η μέρα ψηφοφοριών. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν το χρόνο που σα παρέχετε ώστε να επεξεργαστείτε του συμβιβασμού. Διότι εμεί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν με αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη και περνάμε στο σημείο 8. Δίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μαριαν Χάρκιν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαργής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020 ώστε να μα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής τη. Κυρία Χαρκίν, έχετε το λόγο. Κύριε Λούδιξον. Ναι, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Συνεπώ αναβάλουμε την ψηφοφορία έτσι. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χαρκίν, το σχέδιο γνωμοδότησή σα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη όσον αφορά τη σημερινή μας συνεδρία στο πρωί για τον προπολογισμό. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι υπάρχει μία ε, μειοψηφία που μπλοκάρει τα πάντα στο Συμβούλιο. Το ενδιαφέρον για αυτή τη μειοψηφία όταν είχαμε για παράδειγμα τους Γερμανούς συναδέλφους εδώ περιέγραψαν το EGF ως το μικρότερο από τα προβλήματα, ως το, λάθος, συγγνώμη, το, τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Τα υπουργεία που χρησιμοποίησαν το EGF πολύ συχνά δεν επικοινωνούν με τους, με τους υπουργούς οικονομικών ή δεν συμφωνούν πάντα. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε και αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε με τους δύο συνεισηγητές, τον κύριο Κάλφιν και τον κύριο Μπολγκέρ για το MFF, για το ΔΟΠΟΔΟ. Και ο κύριος Μπολγκέρ ανέφερε κάτι ενδιαφέρον για το EGF, ότι σε αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μια μελέτη όσον αφορά την νομική βάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και θεώρησε ότι έτσι το Συμβούλιο ίσως να μην είναι σε θέση να απορρίψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Είπε επίσης ότι αρχικά είχε αμφιβολίες για αυτό το ταμείο, αλλά τώρα το υποστηρίζει. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ε, Επίση, ο πρόεδρο μου έλεγε μετά τη συνάντηση ότι ίσω να υπάρχει η δυνατότητα η Επιτροπή να ξανεποβάλει το ζήτημα για το 2013 και έχετε μιλήσει και εγώ μιλάω, θα μιλήσετε με την Κυπριακή Προεδρία και θα μιλήσω εγώ και με την Ιρλανδική Προεδρία. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Θα ήθελα επίσης Πρόεδρος να μας το εξηγήσει μετά τη σημερινή συνεδρία. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει το EGF σε κάποιο μηχανισμό αναδιάρθρωσης. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό αργότερα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ζήτημα που μας απασχολεί από την αρχή είναι το ζήτημα της αρμοδιότητας. Αναμένουμε ακόμη μια τελική απάντηση. Πιστεύουμε ότι θα τη λάβουμε στις 20 του μήνα της, έχω μιλήσει με τον κύριο Άλβες που κάνει την γνωμοδότηση στην Άγκρη και δεν έχει συζητήσει αυτό το ζήτημα ο κύριος Άλβες ε, από τότε που ξεκίνησε το ζήτημα εδώ και μήνες. Ενστικτοδός θα έλεγα ότι πιστεύω ότι η Άγκρη θα συμφωνήσει αρκετά με την άποψή μας. Οπότε μπορεί να επιτύχουμε συμφωνία γι' αυτό, αλλά ίσως είναι προτιμότερο να περιμένουμε για να δούμε τι θα πει η Επιτροπή Άγκρη. Τώρα όσον αφορά το ίδιο το σχέδιο έκθεσης. Ε, κάναμε πολλέ ε, συνεδριάσει με τους Κιώδε πριν από αρκετό καιρό. Τότε οι συζητήσεις ε, μου παρήχαν πολλά στοιχεία για τις τροπολογίες που έκανα για αυτό την έκθεση. Επίσης ενημερώθηκα στη συνεδριάση μου με την ΕΟΚΕ, την Επιτροπή των Περιφερειών, την ενδιάμεση αξιολόγηση και τις εκθέσεις ομάδων εργασίας που επισκέφθηκαν διάφορες χώρες και την ομάδα εργασίας EGF για να σας παρουσιάσω τώρα συνοπτικά κάποιες λεπτομέρειες γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω τι έχουν από οι άλλοι παρά αυτά που έχω γράψει εγώ. Εγώ έχω διαγράψει τη νομική βάση, δεν έχω διαγράψει τη λέξη αγρότη σε κάθε περίπτωση. Την έχω αφήσει στην ίδια βάση με τους αυτοαπασχολούμενους, παρότι τα διαφορά μέλη μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, ε, θα ήθελα να τις ακούσω. Ένα από τα επιχειρήματά του να έχουμε τους γεωργούς ε, κάτω από την πρόταση της Κομισιόν είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέπουμε αναδιαρθρώσεις στον ένα τομέα και όχι στον άλλο. Τι γίνεται με την βιομηχανία; για παράδειγμα. Θα ήταν άνηση η αντιμετώπιση. Εγώ συμμετέχω και στην Επιτροπή Γεωργίας, συνεπώς το θεωρώ ότι το μέσο αυτό δεν είναι επαρκές. Θα... Πρέπει να είναι ισότιμο, να αντιμετωπιστεί ισότιμο το ζήτημα. Άλλα ζητήματα που αναφέρω στις τροπολογίες μου είναι οι έγκαιρες δράσεις. Θα ενδιαφερόμουν να μου πει η Κομισιόν τι θεωρεί γι' αυτό. Θα με ενδιαφέραν οι απόψει τη Κομισιόν για αυτό το θέμα. Επίση, η χρηματοδότηση. Αυτό το ζήτημα κατ' κατά επανάληψη. Είναι δίκοπο μαχαίρι, διότι μερικά κράτη-μέλη θέλουν η συγχρηματοδότηση στο 50% και άλλα δεν θα χρησιμοποιήσουν το EGF γιατί η συγχρηματοδότηση δεν είναι αρκετά υψηλή. Το γνωρίζω αυτό μετά από συνομιλίες μου με διαφορούς υπουργού. Προτείνω λοιπόν να έχουμε 50%, 65% για λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και 75% για χώρες ε, που ε, βρίσκονται σε πρόγραμμα διάσωσης ή λαμβάνουν χρηματοδότηση από το EFSF και το καθεξής. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω την άποψη των μελών για αυτές τις προτάσεις. Επίσης ανέφερα στην έκθεση για τις εξαιρέσεις για χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Ένα ζήτημα μου έχει κάνει εντύπωση Κοιτώντα τι διαφορέ αιτήσει που λαμβάνουμε στην ομάδα εργασία EGF, κοιτώντα τις λεπτομέρειε πώς δαπανώνται τα χρήματα και το καθεξής, μία από τις αδυναμίες, ε, θεωρώ κατά την άποψή μου στο EGF, είναι ότι ορισμένες φορές, όχι πάντα, μόνο ορισμένες φορές, ορισμένα κράτη-μέλη σχεδόν χρησιμοποιούν το EGF ε, ως ε, ένα ταμείο εξελισσόμενο και αναρωτιέμαι κατά πόσο αξιοποιείται καταλήλως. Έχουν αυτό που ονομάζεται pecuniary allowance. Σύμφωνα με την νομοθεσία που προτείνεται, ε, οποιαδήποτε επιδόματα που πρότεινα για αυτά τα επιδόματα που χαρακτηρίζονται ε, επιδόματα pecuniary, χρηματοοικονομικές απώλειες ε, όπως έχει σήμερα η ένα μέλος δηλαδή χρηματοδότηση 50% φυσικά χρηματοδοτεί το 50% αυτών των επιδομάτων αλλά πιστεύω ότι για να δώσουμε προστιθέμενη αξία ειδικότερα στους απολυμμένους εργαζομένους λόγω υπερβαλλοντος προσωπικού ή ανέμεναν ότι θα υπήρχε προσθέμενη αξία για τους ίδιους τους εργαζομένους και ίσως αυτό θα ήταν η κατάλληλη οδός. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα γίνει δεκτό από τα κράτη-μέλη τα ίδια, αλλά και πάλι θα με ενδιαφέρει να ακούσω τα σχόλια των μελών. Ένα-δυο τελευταία σχόλια προσπάθησα να ευθυγραμμίσω το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με τους στόχους ε, της Ευρώπης για το 2020 και προσπάθησα να το συμπεριλάβω αυτό στην έκθεση. Ένα σημείο που συνάντησα πολλέ φορέ τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση αλλά και στην επαφή μου με του εργαζομένου είναι ότι υπάρχει ανάγκη να πάσα στιγμή οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους να συμμετέχουν στην ε, σύνταξη του δέσμης μέτρων συντονισμού για τους εργαζομένους. Έχουμε σαφή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν αυτό συμβαίνει. Προσπάθησα λοιπόν να συμπεριλαβώ και αυτό στο κείμενο την ανάγκη εμπλοκή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εκπρόσωπων των εργαζομένων ή του ίδιου του εργαζομένου. Το τελευταίο σημείο επίση αφορά την ανάγκη προορατικής ε, αλληλεπίδρασης ε, μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών. Ορισμένα κρατημέλη βλέπουμε από τις αιτήσει τους είναι πολύ προενεργά και αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Ε, άλλα κρατημέλη χρειάζονται να μάθουν από τις βελτιστές πρακτικές για αυτό το λόγο. Αύξα τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτό. Κανείς φυσικά δεν συμφωνεί με αυξήσεις προϋπολογισμών διότι είναι χρήματα που παίρνουμε από τους εργαζομένους. Αλλά βάσει της εμπειρίας μου με το EGF όσο καλύτερα προετοιμασμένο είναι το πακέτο εξατομικευμένων υπηρεσιών και όσο περισσότερο συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταιροί και οι εργαζόμενοι, τόσο είναι καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για τους εργαζομένους. Γι' αυτό το λόγο προτείνω αυτή την αύξηση. Πιστεύω ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία, κυρία Πρόεδρε, και θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταρντέν και με, ε, κυρία Πουσέ. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες σκέψεις γενικού περιεχομένου όσον αφορά το περιεχόμενο της εκθέσεως. Καταρχήν ευχαριστώ για την απόφαση να ε, καταρτιστεί η έκθεση. Πρέπει ε, λοιπόν να θεωρήσουμε ως καλό ότι υπάρχει αυτή η έκθεση που καταρτίζεται και ασχολείται με το θέμα αυτό ενώ άλλοι ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής αλλά με αρνητικές προθέσεις διότι αναφερθήκαμε από ε, μία επαναλαμβανόμενη μειονότητα, μειοψηφία η οποία μπλοκάρει τις αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα και εδώ μιλάμε ακόμη και για πλήρη κατάργηση αυτού του ταμείου. Οπότε όπως βλέπουμε και εδώ, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ακροάσεως αλλά και τους τελευταίους μήνες, το ταμείο αυτό είναι χρήσιμο και ορισμένες φορές είναι προς όφελος ορισμένων κρατών μελών το, ε, τα οποία το αμφισβητούν και αυτό είναι ε, ε εντυπωσιακό γι' αυτό και με ευχαριστεί η θέση του Επιτρόπου Άντορ που μας το επανέλαβε χθε σχετικά με την αναδιάρθρωση στον τομέα της σιδηρουργίας που είπε ότι στηρίζει αυτή την, αυτό το ταμείο και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι με το μέρος μας σημαίνει ότι... Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα την έκθεση, με τα χαράς διαπιστώνω ότι υπάρχει μία σύγκληση την οποία συζητήσαμε επανειλημμένως ε, πριν την κατάρτιση της εκθέσεως και σύγκληση της ε, εκθέσεως αυτής με τους ε, άλλους ε, εισηγητές θέματα συγκεκριμένα που αναφέρονται ή στη γεωργία διότι μιλήσαμε και για την κατάρτιση των κοινωνικών εταίρων και για άλλα σημαντικά θέματα. Ε, όσον αφορά την έκθεση πέραν ε, των ε, γεωργών υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν, που δεν είναι ο στόχος αυτού του ταμείου αλλά υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις με μόνο δύο-τρεις μισθωτούς οπότε ε, πρέπει ίσως ε, να οριοθετήσουμε τη σχέση ε, επιχειρήσεων και μισθωτών για να ξεχωρίσουμε σε ποιο σημείο ξεκινούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να παρουσιάσουμε όμως πιο σαφώς την ε, πρόταση αυτή πιστεύω ότι θα έπρεπε αναλόγως της ε, καταστάσεως της αγοράς εργασίας στην περιοχή να προσαρμοστεί η σχέση αυτή και το ποσοστό αυτό το οποίο προαναφέραμε. Θεωρούμε όμως ότι η παρούσα συγκυρία είναι μία τροχοπέδη για αυτό το ταμείο, ιδίω το, δηλαδή το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, εγκοσμιοποίηση και βλέπουμε ότι ε, το να υπάρχουν απολύσεις σε προσαρμοσμένο επίπεδο είναι αστείο ε, διότι το συζητάμε και στο θέμα της διακυβέρνησης την ανάλυση των προϋπολογισμών των χωρών θα πρέπει διαφορετικά να λαμβάνουμε υπόψη τις, ε, τις ε, επενδύσεις ε, για θέματα συγχρηματοδοτήσεως και ούτω καθεξής. Ακόμη και αν είναι διαρθρωτικά ταμεία ή ε, ε, ε, διάφορα άλλα. Κάπως πρέπει να οργανωθούμε για να στηρίξουμε τη στρατηγική 2020. Όσον αφορά τις γεωργικές ε, επιχειρήσεις, ε, όταν δεν θα υπάρχει πια μία συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέπει να προωθήσουμε τα προγράμματα τα οποία ενισχύουν την Ευρώπη και να το συνδυάσουμε με τις αναδιαρθρώσεις που θα παρουσιάσει ο Αλεξάνδρος στη συνέχεια. Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει τομεακή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τον τομέα σε κρίση και ε, να υπάρξουν πιο ταχύες διαδικασίες για τις αναγνωρισμένες επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω ότι μία διασύνδεση με την έκθεση που πραγματευτήκαν προηγουμένως ε, είναι σκόπιμη και σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Η κυρία Μωρόν Σορτιέ και μετά η κυρία Κονέλησεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Νάρκιν για το έργο της ε, σε αυτή την έκθεση για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι γνωρίζει πολύ καλά αυτό το θέμα και αυτό το Ταμείο. Ενώ αυτό το Ταμείο γενικά είναι άγνωστο στα κράτη-μέλη. Όχι μόνο στα κράτη, κυρία Πρόεδρε, και εντός του ίδιου μας του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι πρέπει να ε, κάνουμε όλοι μια κοινή προσπάθεια διότι ακούμε πολλές αντιδράσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ενώ κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει καλά την ωφελία του. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ενώ ακόμα πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση με τον Επίτροπο Αντόρ, με, τον Μικαέλ Πορτάς, ο οποίο ήθελε στην εκθεσή του αυτό το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο δεσμευμένο κονδύλιο του προπολογισμού. Και αυτό είχε δεσμευτεί για την στήριξη αυτού του ταμείου, γνώριζε όλη του την εμβέλεια και την επιρροή του και ήθελε να το διατηρήσει και στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε ένα πραγματικό καθήκον να ενώσουμε τι προσπάθειές μα ε, για να διατηρήσουμε και να κάνουμε γνωστό αυτό το ταμείο. Το δεύτερο σημείο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω αφορά να συμφωνήσω με όσα είπε η κυρία Έρκιν για το πόσο κρίμα είναι που δεν επιτύχαμε την εξαίρεση για περιπτώσεις κρίσης και την παράταση της εξαίρεσης για περιπτώσεις κρίσης σε αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτή η απόφαση είναι σκανδαλώδης και ακατανόητη. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να μαχηθούμε ώστε αυτό το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση να μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ή σε πραγματικές συνθήκες κρίσης που επηρεάζουν τους μισθωτούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν όσον αφορά τη θέση της για το άνοιγμα, το προτινόμενο άνοιγμα στον αγροτικό κόσμο. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν έχει σχεδιαστεί υπό αυτό το πνεύμα. Συνεπώς δεν είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα, δεν αποτελεί λύση, επαρκή ευκαιρία Σε αυτό συμφωνούν και οι ειδικοί στη Γεωργία της Κομισιόν θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση οι διεθνείς συμφωνίες να αποσταθεροποιήσουν τόσο πολύ το γεωργικό κόσμο που να χρειάζεται αυτός ε, να καταφύγει στο Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετικού ταμεί και θεωρώ ότι δεν πρέπει να του αναμίξουμε. Το τέταρτο στοιχείο, σημείο για το οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι η αναγκαιότητα εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα πιο πρώιμα στάδια των διαδικασιών που σχετίζονται με το ε, Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε διαπιστώσει ήδη στο παρελθόν, η ιστορία μα το αποδεικνύει και η πραγματικότητα μα αποδείχνει ότι όταν δεν εμπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι, το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση δεν λειτουργεί σωστά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ε, ωφελεί ενδιάμεσου που δεν χρειάζονται καθόλου τη στήριξη αυτού του Ταμείου. Τέλος, ε, δεν συμφωνώ καθόλου με το φίλο μου τον Φρεντερίκ Νταρντέν. Συμβαίνει διαφωνίες και πρέπει να στο πω ειλικρινά. Όσον αφορά τα όσα είπες, για την πρόσβαση του Ταμείου στις, για τις μικροεπιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες. Έχω δει τους φακέλους που έχουν περάσει από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μερικές φορές όταν μιλάμε για μια ε, μικροβιομηχανία, ε, κεραμικής, βιοτεχνία, ε, ξύλου. Έχουμε που επηρεάζεται. Έχουμε ένα δίκτυο μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μερικές φορές με έναν υπάλληλο μισθωτό, που επηρεάζονται σε θέματα υπεργολαβίας. Αντιθέτως, πιστεύω πρέπει να προωθήσουμε την πρόσβαση σε αυτό το ταμείο για βιοτεχνίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι αυτό που επιθυμούμε στο επίπεδο του ΕΛΚ. Πιστεύω ότι πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό. Κυρία Κορνέλισεν και μετά η κυρία Λοπεφοντανιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πολύ καλή δουλειά που έγινε σε αυτό το κείμενο απομένουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια στις γενικές γραμμές. Η εξαίρεση για περιπτώσεις κρίσης και ε, η επαναφορά αυτής της εξαίρεση θεωρώ είναι ζωτική σημασία και πριν το 2014 και θα ήθελα να μας ενημερώσει η Προεδρία για το πώ προχωράμε σε αυτό το μέτωπο. Το να συμπεριληφθούν οι Γεωργοί υπό τις ίδιες συνθήκες πιστεύω είναι δίκαιο. θα σημαίνει ότι πιθανώς δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πολύ, αλλά ανοίγει τις δυνατότητες σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί γεωργοί σε σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια που ταυτόχρονα χάσουν τα αγροκτήματα του λόγω της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης και χρειάζεται επανεκπαίδευση για άλλα επαγγέλματα. Μ' αρέσει ο ισχυρότερο δεσμό με το Europe 2020. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά έχει ελάχιστα χρήματα να ξοδέψει και ό,τι δαπανίσουμε θα πρέπει να επικεντρωθεί στους κύριους στόχους μας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι το EU 2020. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω περαιτέρω με την συγκήτρια και τους υπολείπους σκιώδης πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εντάξουμε το EGF στο EFSF e e ως ταχύ μηχανισμό ενδεχομένως στο πλαίσιο του EFSF θα παρουσίαζε κάποια πλεονεκτήματα συνοχή για την ανάπτυξη ούτως ή άλλως πρόκειται για χρήματα του ESF οι αιτήσει θα μπορούσαν να διεκπαιρώνονται πιο γρήγορα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ίσως αυτός θα είναι ο τρόπος διάσωσης του Ταμείου διότι η πραγματική μάχη δεν θα είναι στην Επιτροπή Άγκρη αλλά στο Συμβούλιο Πολλές χώρες έχουν πρόβλημα με την ανάπτυξη του EGF, ε, πολλές αναφέρονται σε θέματα επικουρικότητας και πολλές φορές δυστυχώς έχουν δίκιο. Αλλά για μας είναι αυτό που είναι σημαντικό είναι τι κάνει στην πραγματικότητα το Ταμείο αυτό. Κάνει τη διαφορά για ανέργους, για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που το χρειαζόνται περισσότερο από όλου. και θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από τα ζητήματα επικουρικότητας, ειδικότερα αν καταφέρουμε να το στοχεύσουμε καλύτερα και να φροντίσουμε να καταλήγουν τα κονδυλιά του εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και όχι να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα για τα πλουσιότερα κράτη-μέλη. Η ενσωμάτωση λοιπόν του EGF με το ESF ίσως να είναι μια λύση. Επίσης η κυρία Χάρκιν να μιλάει για δυνατότητες μετατροπής του σε ταμείων αδιάρθρωσεων. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω περισσότερα και γι' αυτό και ειδικότερα μάλιστα όσον αφορά και το πρασίνισμα, το greening της οικονομίας. Ευχαριστώ η κυρία Λόπες Φοντανιέ και η κυρία Μπλίνκη Μπιτσοτέχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να προσθέσω κάποια πράγματα. Ήθελα να πω ότι υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό την εισηγήτρια. Θεωρώ ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το Ταμείο ώστε να βελτιώσει σε επιλογές απασχολησιμότητας των απολυμένων και ε, ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το σωστό προπολογισμό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις τρέχουσες ε, συνθήκες που εδώ και κάποια χρόνια είναι αρκετά σκληρές. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση της εισηγήτριας όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Θεωρώ ότι αυτά θα βελτιώσουν και θα διευκολύνουν τα πράγματα για τα κράτη-μέλη ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο Ταμείο. Πιστεύω επίσης ότι είναι θετικό σημείο που αυτός ο κανονισμός ε, αποδέχεται ε, ως κριτήριο τις προσωπικές συνθήκες, τις προσωρινές συνθήκες κρίσης ε, και το... όσον αφορά του γεωργού, θεωρώ ότι πρέπει όντω να αντιμετωπίζονται ισότιμα με του υπολείπου εργαζομένου. Και παρότι δεν αναφέρονται ρητά σε μεγάλο κομμάτι του κειμένου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υποθεί καθαρά ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι γεωργοί ισότιμα, το ίδιο και οι πολυπεργαζόμενοι. Αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. Διότι δεν μπορούμε απλά να παραβλέπουμε τους ε, γεωργού. Πρέπει και αυτοί να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Τέλο, ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτω με την Ελιζαμπέτ Μογανσάχτιε. Πιστεύω και το πιστεύει και η Κομισιόν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την προσωρινή εργασία ή τους εποχιακούς εργαζομένους ή και τους εργαζομένους με μόνιμες συμβάσεις αλλά και αυτούς που έχουν προσωρινές συμβάσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις στην Ισπανία. Έχουμε πολλές μικροεπιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς και θεωρώ ότι είναι σημαντικό για αυτές τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο. Κυρία ευχαριστώ. Την, ε, την εισηγήτρια η οποία όντως έκανε μεγάλη προσπάθεια για να καταρτήσει αυτό το έγγραφο και θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια. Στο Συμβούλιο υπάρχει ακόμη μία μειονότητα η οποία μπλοκάρει το θέμα και αυτό οφείλεται σε τη Γερμανία ε, διότι η αρμόδια ε, υπουργό στη Γερμανία εξήγησε ε, πώς ε, αντιλαμβάνεται το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και η άποψη ήταν θετική. Με εκπλήσει λοιπόν τώρα η θέση που εκφράζει στο Συμβούλιο η Γερμανία. Το ερώτημα το οποίο θα ήθελα ίσως να μπορέσω να εξηγήσω στον εαυτό μου είναι ότι εφόσον έχουμε το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και άλλα και ταμεία, εάν τα συγχωνεύσουμε θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Αλλά δεν βλέπω κανένα να ενδιαφέρεται. Οπότε δεν συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Κορνέλησεν η οποία λέει ότι το Ταμείο της Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να συγχωνευτεί στο ε, κοινωνικό ταμείο διότι τότε θα χάναμε πόρους και θεωρώ ότι δεδομένη της κρίσης ε, στο περιβαλλοντολογικό τομέα. Το ταμείο αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα και πρέπει να διατηρηθεί το ταμείο αυτό και να συνεχιστούν οι προσπάθειές του. Ε, συμφωνώ με τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι ε, η ιδέα για την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων εις το Ταμείο Προσαρμογής της Παγκοσμιοποίηση είναι σημαντική. Οι άνεργοι που έχασαν τη δουλειά τους θα έπρεπε να μπορέσουν να αποζημιωθούν και ε, το, οι πόροι δεν είναι επαρκή στα περισσότερα κράτη ε, δεν θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν επικοδομητικά και γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουν σε 75% ε, χρηματοδοτήσεως. Όσον αφορά τη γεωργία, ε, το έχω πει και το ξαναλέω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έμπλεξε σε αυτή την κατάσταση διότι προσπάθησε να βάλει ε, τους 3 ε, εκατομμύρια για τους γεωργούς αλλά χρειαζόμαστε 7 θέλουμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τους γεωργούς ή να τους βοηθήσουμε και ε, θα ήθελα να χρησιμοποιηθούν υπό συγκεκριμένε συνθήκες. Λοιπόν, Είμαι μέλος της ε, Επιτροπής Γυναικών Επιπλέον. Έχουμε ετοιμάσει μία γνωμοδότηση επί του θέματος και θα ήθελα να ζητήσω την, ε, από την εισηγήτρια να λάβει υπόψη σε αυτή την γνωμοδότηση η οποία είναι πολύ σημαντική όπως επίσης η πτυχή των γυναικών και της ισότητας. Ο κύριος Τόμας Μαν, η κυρία, η κυρία μπορώ να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ωραία, τότε ο Τόμας Μαν τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Μάριαν σίγουρα κατάρτισε όπως συνήθως μία καλή έκθεση και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε επικοδομητικά. Αλλά υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία πρέπει να θίξουμε. Κυρία Μπλίνκτσουτούτε, ε, η Γερμανία ε, χρησιμοποιεί την ε, δεσμευτική μειονότητα διότι έχουμε αρνητικές εμπειρίες στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι δεν είναι η τελευταία λέξη της εμείς ε, οι ευρωβουλευτές ε, όμως ε, δεν είναι τόσο μακριά από τις χώρες τους και μπορούν να επέμβουν. Θεωρώ ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση έτσι όπως έχει διατυπωθεί, όπως το επεξεργάστηκε επακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν είπαμε ότι δεν θέλουμε να ξοδεύουμε χρήματα αλλά να είμαστε εστιασμένοι όπου υπάρχουν ανάγκες αυτό δεν έχει αναγνωριστεί περιοριστεί σε ορισμένες ε, πρωτεύουσες ε, και δεν ξέρω αν οι προσπάθειές μας θα είναι ε, επιτυχής για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Επίσης έχουμε τώρα ένα ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, το διακηρύσει πομποδός ο κύριος Βαρόσο και μετά λέει αυτά τα χρήματα θα τα αφαιρέσουμε από το ESF. Ε, e Δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν έτσι. Πρέπει να διαχωρίσουμε τα θέματα και γι' αυτό το Ταμείο για την ε, Παγκοσμιοποίηση έχει αναπτυχθεί, είναι αποτελεσματικό και ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε ένα κορβανά και τον μοιράζουμε όπου χρειάζεται. Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια τα οποία να γίνονται σεβαστά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνονται όλοι. Όσον αφορά την γεωργική πτυχή, ε, έχουμε τη γεωργία που μας ενδιαφέρει και ξέρω ότι όπως και οι συνάδελφοι ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει διότι δεν μπορεί αν ε, έχουμε συγκεκριμένα στη, ε, θέματα για να στηρίξουμε τους γεωργούς που έρχονται από το ΦΕΟΓΑ να αφαιρεθούν ή να περιλάβουμε τους γεωργούς στο Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχουν σωστή θέση εδώ οι γεωργοί στο Ταμείο της της παγκοσμιοποίησης και δεν θα χρησιμοποιηθούν σωστά οι πόροι. Θα δούμε όμως στις τροπολογίες και στις συζητήσεις αν μπορέσει να υπάρξει μία συνενετική αντιμετώπιση αλλά ε, ήθελα απλούστατα εδώ να παρουσιάσω τις θέσεις μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Έχει το λόγο ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ και συμφωνώ με όσα έχουν προταθεί, ούτω ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης του ΦΟΓΑ. Πέρασε ένας χρόνος, έχει αρχίσει αυτή η διαδρομή. Επίσης, συμφωνώ για το ότι από το Ταμείο θα πρέπει να εξαιρεθεί, μάλλον από το περίφημο ταμείο, η Γεωργία. Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί μια εξισορρόπηση μεταξύ κρατικών, εθνικών αρμοδιοτήτων και αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της επικορικότητας. οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υποστήριξη, για τη βοήθεια στις ΜΜΕ είναι οι υπηρεσίες των κρατών μελών. Και θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να βοηθάτε ο, ο, όλος ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητα. Αν τώρα έχουμε κάποιες ΜΜΕ με έναν ή δύο μόνο εργαζομένους, τότε αυτό είναι θέμα, δεν είναι θέμα πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών παρόλα αυτά. Έχουμε ακόμα κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να, να γίνουν. Ε, και θέλω τώρα να σας πω για περσιμία ότι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, ξέρετε ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής είχε απασχολήσει την Ιδανέζικη Προεδρία. Και είχε πει η Ιδανέζικη Προεδρία ότι μετά το 2014 δεν θα λειτουργεί. Όλοι εδώ, πεπισμένοι, είμαστε για την χρησιμότητα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Έχουμε και το Συμβούλιο το οποίο θα γίνει αύριο, θα γίνει για την επόμενη εβδομάδα, ε, το Ταμείο Γενικών Υποθέσεων, οπότε οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. παντός επί της ε, ουσίας έχουμε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι θέμα απλά σύμφωνη γνώμη. Δεύτερον, η εισηγήτρια ε, έδειξε και το ζήτημα του να έρθουν συμβαθεί με το Συμβούλιο για τη συζήτηση που έγινε χθες. Για το τι θα κάνει η Κυπριακή Προεδρία. Σήμερα στο Συμβούλιο συζητείται η πρόταση της παράτασης της εργαστή της ισχύω της υπάρξεως του Ταμείου Προσαρμογής. Από το 2012-2013 γιατί καταρχήν είχε προβλεφθεί για μία μικρή περίοδο και είχαμε πει ότι 31 12 του 2011 θα πάψει να λειτουργεί στο Δεσυμβούλιο προσθέθηκαν χρόνια και, και ήταν τέλο πάντων 2012, πάει το 2012. Θα ήταν ε, άσχημο το να αποσύρει η Κομισιόν την πρότασή τη. Οπότε τώρα την τροποποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι τώρα σας κάνουμε πρόταση και θα αποφασίσετε το 2013 μια που δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Συμβούλιο, αλλά αν θέλουμε να στείλουμε ένα σωστό μήνυμα, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το τι θα γίνει με την ε, Επιτροπή Γεωργίας. Ελπίζω ότι τελικά θα έχουμε συμφωνία σε σχέση με την κατανομή των αρμοδιοτήτων Μας είπε και η συγκήτρια ότι επί της ουσίας μέσα στο ίδιο μήκος κύματος. Πάντως, για να δούμε τα, τα δύο βασικά σημεία αυτής της έκθεσης πρώτα-πρώτα. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν. Είναι απαράδεκτη. Κάτι γνώμη μας. Νομίζω ότι είναι στοιχείο με το οποίο θέλουν να καθησυχάσουν κάποιες χώρες σε σχέση με την αλλαγή στην ερωτική πολιτική, να τους καλοπιάσουν ότι δίθεν ε, νοιάζουν για τους εργάτες. Άρα δεν μας αρέσει για αυτό το λόγο, αλλά δεν μας αρέσει για κάποιο άλλο λόγο η πρόταση της Κομισιόν, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες των συμφωνιών για τις ελεύθερες συναλλαγές. Μα είναι να έχουν τέτοιες επιπτώσεις, τότε θα έπρεπε αυτές οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών να έχουν λάβει άλλη μορφή. Αλλιώς να σηκώσουμε τα χέρια, να πούμε ωραία, κάντε ό,τι συμφωνία θέλετε και να ξεχάσουμε τους, ε, τους γεωργούς. Είναι το αντίθετο του είναι το αντίθετο της αηφόρου ανάπτυξη. Όλα τα αντίθετα. Ε, σαν να ενθαρρύνουμε την, ε, την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος, σαν να θέλουμε να τιμωρήσουμε τις χώρες αντί να τις βοηθήσουμε, τις τρίτες. Και στην ομάδα εργασίας Θυμάμαι, υπήρχε μια περίπτωση στην Ισπανία που είχαμε πόσες, πόσους 500 επιχείρησεις. Θυμάμαι ακριβώ. η Ισπανική Προεδρία ήθελε να συζητηθεί το θέμα της κοινωνικής προστασίας των ελευθέρων επαγγελματιών σε συγκυρία κρίσης. αυτοί που δεν δικαιούνται επίδομα ενεργείας, άλλο επίδομα πρόνοιας και βρίσκονται ξεκρέμαστοι. Οπότε το να ληφθούν υπόψη αυτές οι περιπτώσεις οι ατομικές που να καλυφθούν όπως και για κάποιους ε, γεωργούς είναι μια σκέψη ενδιαφέρουσα, κάτι άλλο. Η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν ξέρω που θα πάει το θέμα, αλλά αν θέλουμε το Ταμείο Προσαρμογής να κινητοποιείται πιο γρήγορα, κάτι το θέλουμε όλοι, θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα για τον προπολογισμό. Γιατί η σημερινή δημοσιονομική κατάσταση εξηγεί τι έγινε. Ε, αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης που παίρνει τόσο, τόσο, τόσο χρόνο αυτά και τώρα για την εισηγήτρια, κάτι που είπε είναι αλήθεια ότι το είπαμε πολλές φορές για αυτή την συνάρθρωση που είπε ο κύριος Νταρντέν για το Ταμείο Προσωπικής Παγκοσμιοποίηση και αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεση ΣΕΡΚΑΣ, πρόκειται για κάποιες προτάσεις που ε, ξεκίνησαν με γαλλική πρωτοβουλία, αξίζει να τα εξετάσει κανείς καλύτερα Το πώς σε αυτό το Ταμείο Προσαρμογής θα μας οδηγήσει σε καλύτερη αναδιάρθρωση. Αυτά είχα να σας πω και τώρα πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Περβάν σε ένα σύντομο σχόλιο για αυτό το ζήτημα που ανέφερες εδώ. Ε, πιστεύω Τώρα θα ήταν πρόβλημα να το αναμίξουμε αυτό διότι το ESF κατανέμεται σε εθνικό επίπεδο, σε επιχειρησιακά προγράμματα, είναι ένα διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία παρότι εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο τη βοήθεια στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης Καλό θα ήταν να μην τα αναμίξουμε, θα ήταν επικίνδυνο. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω την κυρία Χάρκη να μην τα παρατήσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα ήθελα να πω ότι θα σας υποστηρίξουμε σε αυτή τη μάχη. Έχει αλλάξει η μορφή η κρίση σε μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρειάζεται πια Απλά λέω ότι αν δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές που θα το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό. Είναι απολύτως σαφές ότι θα πρέπει να κινητοποιείται γρήγορα, θα πρέπει να είναι στοχευμένο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια έκφραση ελληνικής με διαφορετικό όμως τρόπο από ό,τι εκφράζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ είναι το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν οι γεωργοί ή όχι. Εάν οι γεωργοί χρειάζονται κάτι, όπως ε, οι γεωργοί που είναι θύματα της πτώχευσης εταιριών και της κρίσης, και τότε θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ε, ώστε να χρησιμοποιήσουμε ένα ξεχωριστό ταμείο. Αλλά δεν θα χρησιμοποιούσα το EGF για τους γεωργούς. Ε, δεν έχει νόημα να δεσμεύσουμε κάποια ποσά από αυτό για τους γεωργούς. Ε, ίσως να μην είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των γεωργών. Κυρία Προντίνσκι, για την Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την συγκεντρία για την έκθεσή τη. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει και φαίνεται ότι αναζήτησε συνένεση. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η συζήτηση. Βλέπω ότι όλο ο κόσμος θέλει να υποστηρίξει την εισηγήτρια στην προσπάθειά της να βρει μια λύση ισορροπημένη Για του γεωργού, συμφωνούμε όλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα και η έκθεση επίση έτσι όπως ε, έχει παρουσιαστεί είναι πολύ λογική σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να περιλαβούμε και αυτού και του γεωργού όπως και άλλο κόσμο ως επιλέξιμους για ενίσχυση από το Ταμείο. Όμως, αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο είναι αυτές οι πιο λεπτομεριακές ρυθμίσεις, οι αλλαγές, προσαρμογές που έκανε η συγκέντρια στη δική μας πρόταση. Τα περισσότερα πόσα λέει είναι θετικά, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μας. Και εάν τα δούμε λοιπόν ένα προς ένα, θα διαπιστάσουμε ότι, για παράδειγμα, αναφέρεται εδώ ο ρυθμός επανένταξης στο τέλος της περίοδου εφαρμογής και όχι μετά από ένα χρόνο. Λογικό, ε, γιατί έτσι πάμε για δύο χρόνια υποστήριξη από το Ταμείο και πάρα πολλοί από του εργαζομένου πρόκειται να συμμετάξουν σε κάποια προγράμματα τα οποία θα πάρουν δύο χρόνια ή και παραπάνω. Ανάλογα το πότε αρχίζει το πρόγραμμα. Επομένω, είναι λογικό να μετρηθεί αυτή, αυτό το ρυθμό τη πανένταξη στο τέλο τη περίοδου εφαρμογή και όχι ενδιάμεσα. Κάτι άλλο τώρα, το οποίο έχω σημειώσει. Αυτέ οι ενισχύσει επενδύσεων δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 25.000 ευρώ και όχι 35. Νομίζω ότι εάν οι γεωργοί δεν καλύπτονται όπως εμείς στην αρχή είπαμε για τα 25.000 ευρώ θα αρκούν. Και έτσι οι πόροι θα καλύψουν αρκετούς πολλούς εργαζομένους. Μέχρι σήμερα δεν νομίζω το Ταμείο έχει υπερβεί τα 25.000. Επομένω, βολεύει αυτό το ποσό τώρα. Όσον αφορά την τεχνική αρρωγή και το πιο εντατικό ρυθμό τη σε σχέση με την οροφή του 7% και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι η ρύθμιση είναι εύστοχη διότι όπως είπε η συγκεντρία πολλές φορές στην αρχική εφαρμογή από ένα κράτος μέλος πάμε πάνω από το σύνηθες 4% που είναι ο κανόνας. Επίσης, μπορεί να είναι παραπάνω το, το ποσοστό σε κάποιες αμαγρισμένες περιοχές. ή σε περίπτωση ενισχυμένων ελέγχων αν χρειαστούν. Και όσον αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και εν προκειμένου τα πράγματα είναι χρήσιμα αυτά και είναι, είναι θετική και αυτή η ιδέα. Ναι, ναι, Πρόεδρε, ξέρω, θέλετε να μην γρηγορήσω και να σας πω πάρα πολύ σύντομα αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Πρώτη, η συγκεντρία ότι σε περίπτωση και το εκπαίδευση η περίπτωση εφαρμογή μπορεί να αυξηθεί. Αυτό ίσως δεν είναι αυτονόητο πώς θα γίνει, γιατί είχαμε πει για 24 μήνε συν 6. Άρα αυτό ίσως θα πρέπει να συζητήσει λεπτομέρειες του στο πώς θα γίνει τελικά τώρα όσον αφορά την ετησία έκθεση. Από ό,τι μας λένε σήμερα, ότι θα να πάμε για εκθέσεις ανά διετία για εξοικονόμηση ε, προσπάθειας. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο τρομερό. Νομίζω πάντως ότι κάλυψα τα περισσότερα από αυτά που θέλατε και βέβαια, αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Πριν αρχίσω να σας πω για πόση ώρα, δύο ή επτά. Δύο, δύο, δύο λεπτά. Δύο λεπτά, καλύτερα λέει πρώτος. Καλά, καλά, Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προφτάσω, αλλά θα σας τα πω για στον κύριο Νταρντέν και στους άλλους ε, ε, μας είπαν για τις μικρές εταιρείε και μας είπαν ότι εδώ πέρα υπάρχει ε, ένα διαχωρισμό παρολεπτός και όπω ήδη έχετε πει Προ το παρόν έχουμε, έχουμε κάλυψη των μικροεπιχειρήσεων με έναν, δύο, δύο-τρει εργαζομένου και έχουμε και τι και αυτό η ίδια που μας λαμβάνει η χώρα Διάκουσα αυτό το οποίο είπε ο κύριο Νταρντέν και θα το συζητήσουμε τώρα όσον αφορά τον αριθμό συγχρηματοδότηση, Μα είπε ο κύριο Νταρντέν ε, τι γίνεται με την περιφέρεια, τι γίνεται με την αγορά εργασία, πώ έχει κατάσταση και ότι θα πρέπει αυτά να τα δούμε ανά περίπτωση. Ε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο ότι το κάνουμε ε, αλλά είμαι ανοιχτή να το συζητήσουμε. Ε, Επίση, άκουσα Ε, γιατί είπατε για τον κύριο Πόρτας ε, συνάδελφοι, ε, τα ξέρω αυτά που είπατε ε, και βεβαίω και θα ήθελα να υπάρχει αυτή η παρέκκληση για λόγω της κρίσης. Μα υπάρχουν τα, τα, τα υπάρχουν πόροι, το είπανε πολλοί τώρα όσον αφορά τους Γεωργούς, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς. Να καλύψουμε όχι μόνο τους ε, αλλά και όσους μπορούν να εξισωθούν με αυτούς λόγω των συνθήκων μας είπατε κύριε Κορνέλησεν για το Ταμείο Σομονίξης και το Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει πρόβλημα, έχω ακούσει παρατηρήσεις ε, από πολλοί κόσμο να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Πάντως κατά τη γνώμη μου, θα δούμε αν μπορούμε να το, να το κάνουμε έτσι. Βέβαια δεν λέω όχι από τώρα. Μας είπατε για την συγχρηματοδότηση και για αυτά τα επιδόματα είπατε επίσης για την εμποδίουσα μειοψηφία. Όχι, δεν πρόκειται μόνο για τη Γερμανία και είναι και άλλες χώρες. Και μικρές. Γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι αρκετός αυτός ο ρυθμός συγχρηματοδότηση. Ο καθένας μπλοκάρει την απόφαση για τους λόγους του. στο επεξηγηματικό σημείωμα θα τα πω. Πολλές χώρες μέλη ελπίζουμε να αρχίσουν την κάλυψη των μέτρων, να τα χρηματοδοτήσουν, ακόμα και αν είναι σε δυσκολίες, τουλάχιστον έστω εν μέρη. Τέλος, για όσο επί κομισιόν, ευχαριστώ για σε πω μόνο δύο. Όσον αφορά την ενίσχυση επενδύσεις, με, με αρέσει το 25.000 γιατί έκανα έναν υπολογισμό σε σχέση με το πόσο πόσα χρήματα υπάρχουν και είδα τι έγινε μέχρι σήμερα και αν για τις 35.000 θα ήταν υπερβολικό να το αφήσουμε εκεί το ποσό τέλος. Να εξαθέσουμε κάτι για αυτή την διετία. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία αν κάποιος υποβάλει αίτηση για Οκτώβριο-Νοέμβριο προς το Ταμείο Προσαρμογής και κάποιος εργαζόμενος φτάσει στο τρίτο επίπεδο, συνήθως αυτό γίνεται τον επόμενο Σεπτέμβριο σε σχέση με την αφετηρία. Άρα πρόσβαση στην επόμενη ευκαιρία Έτσι θα γίνει σύμφωνα με την Επιτροπή και άρα διμερώ να δούμε την Επιτροπή πόσο στην πράξη θα ρυθμιστεί αυτό. Ευχαρίστω όποιο άλλο θέλει και ο ή απλώ οποιοδήποτε συνάδελφο μπορεί να έρθει να με βρει πρόεδρο. Από ό,τι βλέπω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μακρηγόρησε, αλλά δεν είπε τίποτα όσον αφορά την πρόταση του να επαναδιατυπωθεί η πρόταση τη παράταση ισχύω του συστήματο, του, του, του, του Ταμείου Προσαρμογή Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να ε, αξιοποιήσει αυτή την πρόταση που μου φαίνεται εξαιρετικά ωφέλιμη σε πολλά επίπεδα. Βάσει αυτών λοιπόν έχουμε τώρα προθεσμία 9 Ιουλίου για την υποβολή τροπολογιών στις 12 η ώρα. Φτάνουμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης όπου θα εξετάσουμε την στροπολογίες του σχεδίου έκθεσης της κυρίας Ελιζαμπέτ Μόρα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού του 2006. κυρία Μόρα, η κυρία Μόρα έχει λάβει 426 τροπολογίες δεν την καλώ να τη σχολιάσει όλες, αλλά να μας δώσει μια γενική εικόνα πάνω στην οποία θα συζητήσουμε. Κάνα πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω κυρία Πρόεδρε, κάποια στιγμή αναρωτηθήκατε για αυτή την ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πιστεύω ότι σήμερα όλη η Επιτροπή Απασχόλησης αποκομίζει τα αποτελέσματα του πνεύματος συνεργασίας και της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ όλων των μελών αυτή της ομάδας εργασίας από όλες τις πολιτικές ομάδες. Επιθυμώ λοιπόν καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης που εργάζονται για αυτή την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με ένα εξαίρετο πνεύμα συνεργασίας εδώ και πολύ πολύ καιρό. Αυτό μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε πολύ περισσότερο την εργασία μας Αφετέρου, μας επιτρέπει επίσης ε, να εντοπίσουμε τις πραγματικές ευθύνες της δικής μας Επιτροπής σε σχέση με άλλες ε, Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα εντάχει, επειδή όπως είπατε είχαμε πάνω από 420 τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες, θα ήθελα λοιπόν εντάχει να σας πω να σας περιγράψω το πνεύμα και τις αρχές που διέπουν την εργασία μας. Η αρχή που διέπει την εργασία μας είναι να διατηρήσουμε το κείμενο πλαίσιο και στα εκτιμώντας να συμπεριλάβουμε όλες τις τροπολογίες που αφορούν τον τρόπο υλοποίηση αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ώστε να διαφυλάξουμε, θα έλεγα, την καθαρότητα του κειμένου και την ευκολία εφαρμογής του. Το δεύτερο σημείο που θέλουμε να διατηρήσουμε πολύ ευανάγνωστος τους θεματικούς στόχους και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης μέσα σε μια λογική διατήρησης των ενιών της κινητικότητας, της απασχόλησης, της ε, διαβίωκμάθησης, της καταπολέμησης της στόχιας και της διοικητικής και της αποτελεσματικότητας των ε, κρατικών διοικήσεων. Τρίτη μας αρχή είναι να αποφύγουμε να είμαστε περιοριστικοί ώστε να υπάρχει περιθώριο υλοποίησης για τα κράτη-μέλη. Για ποιο λόγο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο από τη σήμερα, να είναι πιο αποτελεσματικό δηλαδή και η αρχή λειτουργίας μας αποσκοπεί στο να διευκολύνει αυτή τη χρήση από τα κράτη-μέλη. Αυτές οι αρχές ε, παρουσιάστηκαν τώρα και θα ήθελα να αναφερθώ στα σημεία συμφωνούμε, συζητάμε για τα οποία έχουμε λάβει ε, ε, τροπολογίες και για τα οποία θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμβιβασμούς. Αυτή η αρχή του 25% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Συζητάμε από σήμερα το πρωί. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα από όλους τους συμβιβασμούς και τις τροπολογίες. Το δεύτερο σημείο, και αυτό θα συζητηθεί αρκετά, γιατί κάποιες πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν, το 20% δέσμευση του 20% για την καταπολέμηση της φτώχειας, του 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό όσον αφορά τα ποσοστά. Ο δεύτερος μεγάλος άξονας είναι η αντίθεση στη ρήτρα μακροοικονομικής αρεσιμότητας. Δεν θα επανέλθουμε, όλοι συμφωνούμε σε αυτό το τρίτο σημείο. Αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Τέσσερα προβλέπονται στο αρχικό κείμενο, μπορούμε να τα πάμε στα έξι, ώστε να υπάρχει το περιθώριο υλοποίηση. Να διευκολυνθεί η υλοποίηση. Το πέμπτο σημείο είναι η συμπερίληψη των ανειδίκευτων νέων όπως έχουν εξέλθει από τα συστήματα κατάρτισης και θέμα στο οποίο θα πρέπει φυσικά να επικεντρωθούμε. Στις τροπολογίες προσθέτουμε την ένταξη των κοινωνικών εταίρων για τους ίδιους λόγους που είπα και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προηγουμένως, διότι αυτό αποτελεί εγγύηση συλλογική εργασία και αποτελεσματικότητα για το μέλλον. Επίσης επιθυμούμε να εργαστούμε πιο εντατικά σε, μια συλλογική, σε ένα συλλογικό όραμα όσον αφορά την εξέλιξη των ε, θέσεων εργασίας εντός των επιχειρήσεων και συνεπώς την εξέλιξη των ικανοτήτων των μισθωτών στο πλαίσιο της διαβίου εκμάθησης και επικύρωσης των κεκτημένων γνώσεων. Το σύνολο των τροπολογιών επικεντρώνονται σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Σας ανέφερα τις αρχές, τα κυριότερα θέματα και τώρα θα ήθελα να σας περιγράψω τη μέθοδο εργασίας και το ημερολόγιο μας. Βάσει όλων των τροπολογιών έχουμε ήδη από χθε σε μια μεγάλη συνεδρίαση εργασία συλλογική με όλους τους κοιόδης έχουμε ξεκινήσει την εξέταση αυτών των τροπολογιών διότι έχω ήδη εγώ προτείνει καμιά εξενταριά συμβιβαστικέ να μπορέσουμε μεταξύ μας και με όλες τις πολιτικές ομάδες να συνεργαστούμε ώστε να εξετάσουμε, να εντοπίσουμε τα σημεία σύγκλησης βάσει των οποίων μπορούμε να οικοδομήσουμε το έργο μας. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε θα συγκεντρώσουμε τα σχόλια από τα αποτέλεσμα των εργασιών των διαφόρων πολιτικών ομάδων για ε, 3η 26 Ιουνίου 9 ναι, η ώρα το πρωί δεσμεύομαι να συγκεντρώσω όλες τις απόψεις των διαφορετικών πολιτικών ομάδων έως την Παρασκευή το πρωί της ίδιας εβδομάδα, ώστε οι σκιώδεις εισηγητές να έχουν ξανά την ευκαιρία να δουν τις συμβιβαστικές τροπολογίες ώστε και πάλι να μελετήσουμε Τρίτη και Τετάρτη της εβδομάδας του Στρασβούργου, δηλαδή 3 και 4 Ιουλίου έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε όλοι, να συμφωνήσουμε όλοι και ελπίζω χωρίς προβλήματα για την ψηφοφορία της 5 Ιουλίου έτσι ελπίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα από ότι αν χρειαζόταν να ψηφίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων σχεδόν από όλες τις ομάδες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτό το πνεύμα μέχρι την ψηφοφορία της 5ης Ιουλίου. Ευχαριστώ, κυρία Κίνγκαν Κίνγκα Κούτς και ο κύριος Κοσλόφσκι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά και πάλι έχουμε άπειρες τροπολογίες εισηγήτρια όπως είπατε και εσεί στην εισαγωγή σα όμω κατά κάποιο τρόπο έχουμε αυτή την ομάδα εργασία ε, πάρα πολύ χρήσιμη, δούλεψε όλη τη χρονιά και αν αντάλλαξαμε απόψεις, τα είπαμε και δεν αρχίσαμε από το α. Και έτσι τώρα καταλήξαμε σε αυτές τις τροπολογίε γιατί τώρα το βασικότερο μας πρόβλημα είναι οι προθεσμοί που είναι πολύ κοντινοί αν θέλουμε να ψηφίσουμε στις 5 εβδόμου και ταυτόχρονα για ε, τις διατάξεις πλαίσιο που είναι λογικό όποτε και θα πρέπει να επιταχύνουμε τον ρυθμό εργασία. Και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Με τις να, να βελτιώσουμε, να μην χειροτερέψουμε το αρχικό κείμενο. Το αρχικό κείμενο αλλά και πρώτη Κομισιόν είναι αξιόλογα. Πάντως, στα πιο βασικά συμφωνούμε. Ούτε διαπιστώνω υπάρχει κανένα είδου πρόβλημα. Ε, συμφωνήσαμε στα πιο βασικά. Και Αντιστοίχως, να εξεργαζόμαστε τις συμβαστικέ τροπολογίε. Όπως σα είπα, και εγώ τώρα προσπαθώ να μελετήσω του θεματικούς στόχους, ε, αντικείμενο και πολλών τροπολογιών, από πολλέ πλευρέ, οπότε ίσω τελικά χρειαστεί να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτές τις θεματικές ενότητες ανάλογα με το τι απασχολεί το κάθε κάποιος μέλος άρα προσοχή τώρα με τις μικροαλλαγές να μην ε, στενέψουμε τα περιθώρια τέσσερις, άντε έξι τέτοιες θεματικές ενότητες να έχουμε ό,τι είναι πιο σημαντικό. Επίσης, από την αρχή είπαμε ότι θα διαλέξουμε τις πιο σημαντικές και θεματικές ενότητες να το στείλουμε σχετικά με τις εταιρικές συμβάσεις, πώς θα έχουμε κάποια επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα συγκεράζονται τα οποία θα είναι συμβατά με τα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση. Τι εθνικέ στρατηγικέ τέλο πάντων για να έχουμε τελικά αποτελεσματική χρήση των πόρων. Οπότε γι' αυτό και επιταχύναμε το ρυθμό εργασιών όπως τα είπε και η κυρία εισηγήτρια. Έχουμε κάνει ήδη δύο ραντεβού για να τα πούμε. Νομίζω οι πιθανότητε είναι πάρα πολλέ να καταλήξουμε σε κάτι που θα βρίσκει, αν όχι όλε τι περισσότερε τι πολιτικέ πτέρυγε. Monsieur Κοσλοφσκή πήμε να Markin. Dziękuję Pani Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Συγγήτρια η οποία συνέταξε ένα καταπληκτικό κείμενο με πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και κατάλληλες στοχευμένες προτάσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ιδέες που αποτελούν και θέματα των τροπολογιών μου. Θα πρέπει, πιστεύω, να συντονίσουμε περισσότερο τα κοινωτικά μέσα. Ε, θα πρέπει να οριοθετήσουμε με σαφήνεια τις γραμμές που χωρίζουν το μέσο για την καινοτομία του Εράσμους για όλους και το EDF, ώστε να μην επικαλύπτονται, να μην διπλασιάζονται οι προσπάθειες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε συνέργεια. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να προσανατολιστεί προς αποτελέσματα και όχι διαδικασίες. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτό που προτείνει η Κομισιόν, δηλαδή η απλούστευση, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άποψη. Τα καταποκοπήν ποσά, όλες αυτές οι ιδέες που απλοποιούν τις διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράξουν αυτές τις ευκαιρίες και όχι να περιπλέκουν πέραν του δέοντος τις ε, ε διαδικασίες. Ο κύριος Τόμας um, ε, Συγγνώμη. Κυρία Χάρκιν, συγγνώμη, θα μιλήσω εκ μέρου τη Νάντια που δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Είναι πεπισμένη ότι μετά τι επικοδομητικέ διαπραγματεύσει χθε οι περισσότερα σχέδια συμβασμών είναι ικανοποιητικά. Η επικέντρωση στην ορατότητα και την αποτελεσμότητα του ESF είναι πολύ σημαντική. Θέλει να τονίσει ότι πέρα των κοινωνικών εταίρων, οι αρμόδιε τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ καθώ και οι. Ε, γενικότερε ενώσει σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εμπλακούν όχι μόνο στην υλοποίηση αλλά και στην παρακολούθηση και εξολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επίση, θεωρεί ότι οι μετανάστε και οι επιζητούντε άσυλο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ESF. Επίση, μειονεκτώσει ομάδε όπω άτομα που ζητούν άσυλο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το ESF. Τέλο, η Νάντια θα ήθελε να ευχαριστήσει ε, την για την εξαιρετική συνεργασία και για την εκθέσή τη ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία Μακιντέρ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ότι υπάρχει μία ομοφωνία σχετικά με την έκθεση αυτή την οποία θεωρώ εξαιρετική και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Αυτό που θεωρώ επίσης πολύ βασικό ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ότι είναι μια ιστορία επιτυχίας παρόλες τις δυσκολίες διότι πολλά κράτη λέγουν γιατί ε, δεν πάει πιο γρήγορα, γιατί δεν είναι πιο εύκολο. Πολλές, ε, πολλές από τη, πολλά από τα παράπονα είναι αιτιολογημένα. Καλύτερα να είχαμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση αλλά πιστεύω ότι γενικώ το ταμείο αυτό έχει μία προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, αλλά εμείς το βλέπουμε και τα κράτη το αντιλαμβάνονται, διότι μπορούμε να καταλήξουμε στους αποδέκτες πολύ πιο γρήγορα και να υποφεληθούν. Έχω κάνει ε, ορισμένες... Ε, ορισμένες ε, τροπολογίες ε, σχετικά με ε, τα αθλήματα ευρείας συμμετοχής. Βλέπετε τώρα με το ευρώ, ότι, με το ποδόσφαιρο, ότι έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές με τεράστιες αμοιβέ, αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός ευρείας συμμετοχής είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εμπλακούμε. Έχω και συναδέλφους οι οποίοι συμφωνούν και λέγουν ότι πρέπει και αυτό να συμπεριληφθεί διότι διαφορετικά όλο και κάποια ομάδα, όλο και κάποια μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας μένει παραμελημένη και δεν θα είχαμε διαφορετικά τη δυνατότητα να την προωθήσουμε. Άρα θα μπορούσαμε έτσι να επεκτείνουμε τις χρήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μωρέ Σοντιέ, Σοντιέ. Έδειξε πνεύμα σε εργασίες προς όλους τους σιώδες ηγητές. Και, κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να σας επαναλάβω ότι όλοι είμαστε υπέρ του κοινωνικού ταμείου Έχω δει στην πράξη, στην περιφερειά μου, πώς δουλεύει, πόσο βοήθησε τους νέους να μπουν σε αγορά εργασία. Δύο σκέψεις μου, πρώτα πρώτα. Να μην έχουμε επικαλύψεις. Να μην ξαναχρηματοδοτήσουμε πράγματα που χρηματοδοτούνται. Ας πούμε, τα πολιτιστικά. Τα πολιτιστικά να από αλλού, είναι θέμα επιτροπή ε, πολιτισμού, από το αποφύγουμε. Επίση, σύμφωνα με αυτό που είπε η Κίνγκα, για το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε είχαμε πάρα πολύ μικρή συζήτηση σε σχέση με τη λίστα πραγμάτων που πρόκειται να βάλουμε και πολλέ φορέ όμω λείπουν κάποια δέοντα από αυτέ τι λίστες. Προσοχή. Επίσης, ε, να σας πω για κάποιες τροπολογίες δικές μου, για το άρθρο 2, παράγραφος 1 και για το άρθρο 3, 1C. Εκεί που ε, αναζητώ κάποιες ε, απαλληθές. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. Όμως εμείς το βλέπουμε όχι σαν αρχικό στόχο, αλλά σαν αποτέλεσμα της δουλειάς του Ταμείου. Άρα αυτός ο στόχος θα πρέπει να σχεδιστεί με την αγορά εργασίας σαν αποτέλεσμα των όσων κάνουμε σήμερα για την κατάρτιση. Και σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει επανένταξη, ηρωνική κλπ. 164 ή 162 είναι η νομική βάση που εξηγεί πολλά ε, για το που το πάμε και επίσης έχουμε και τους άλλους στόχους του κοινωνικού ταμείου που κατατείνουν στους ίδιους σκοπούς, το λαμβάνουμε υπόψη. Τώρα επίσης ε, πάρα πολύ σύντομα δύο παρατηρήσει ακόμη. Έχουμε ένα ε, ε, κάποιο κείμενο εκεί που αναφέρεται η ισότητα στην αμοιβή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε, να λέμε πάντα ίση αμοιβή για ίση εργασία. Και αυτό βγήκε σε άλλη εκθέση σήμερα. Οπότε φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνείτε. Η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Γιατί άμα λέμε σκέτο ίση αμοιβή για γυναίκε και άντρε, αυτό είναι κάτι που δεν και σύμφωνοι. Τώρα κάτι άλλο το οποίο θέλω να σκεφτείτε είναι το θέμα των ετούντων άσυλο. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων στους οποίους έχει χορηγηθεί άσυλο και εκείνους τους ετούντες οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ε, λάβει την έγκριση της αίτησης. Ναι, επομένως στην πρώτη κατηγορία, αλλά στη δεύτερη όχι. Ε, δεν, δεν δεχόμαστε τη διατύπωση, το σκέτο ετούντες άσυλο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Συγγήτρια. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, δυστυχώς. Την ίδια τύχη δυστυχώς και, και η κυρία Χάρκιν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους Κιώδης, για τη συμβολή τους σε αυτή την έκθεση. Σημείωσα τις παρατηρήσεις. Είμαι βέβαιη ότι θα επιτύχουμε τρόπους διατύπωσης που θα ικανοποιούν όλες τις ομάδες στο μέγιστο και στους οποίους θα εντάξουμε τα ερωτήματα όλων. Θα μεριμνήσουμε ώστε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να επικεντρωθεί στην επαγγελματική ένταξη. Όπως καταλαβαίνω, η επαγγελματική ένταξη αποτελεί σκαλοπάτι για την κοινωνική ένταξη. Και όσον αφορά την ερώτηση του Τόμας Μαν, βλέπουμε καλά ότι όσον αφορά αυτή την επαγγελματική ένταξη μπορούμε να έχουμε περιθώρια λιγμών που επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε πιο διευρυμένα προγράμματα. Κυρία γραμμή μας είναι η επαγγελματική ένταξη χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο δεν σας έχω μιλήσει και το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα. Είναι η ένταξη των εκθέσεων γνωμοδότησης ε, στην εργασία μας. Αυτό θα λάβει η χώρα και θα κοινοποιήσω τις πληροφορίες στο σύνολο των συναδέλφων αυτής της ομάδας εργασίας ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να συνεργαστούν με τις πολιτικές τους ομάδες. Αφού καταφέραμε να είμαστε τόσο γρήγοροι στην εργασία μας μέχρι αυτό το σημείο, και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει μέχρι τις 5 Ιουλίου. Το κείμενο της Κομισιόν ήταν ήδη εξαιρετικά ενδιαφέρον και θετικό και μας διευκόλυνε στη μελέτη. Ε, προχωρήσαμε έτσι και χάρη στη συνεργασία όλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα προχωρήσουμε επιταχύνοντας, Πρόεδρος. Επειδή βλέπω στο ημερολόγιο ότι δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε εκ νέου τις τροπολογίες, ε, τις συμβιβαστικές, ε, ξέρω ότι ε, διάφορα άλλα μέλη της Επιτροπής θα ενδιαφέρονταν να εξετάσουν αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Πότε θα είναι αυτές οι συμβιβαστικές τροπολογίες διαθέσιμες για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπορείτε να μου δώσετε μια ένδειξη για αυτό το σημείο. Κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως προχωράνε οι εργασίες, αυτή τη στιγμή σκιώδεις εισηγητές που εργάζονται σε κάθε πολιτική ομάδα και μελετούν αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ε, συλλέξουμε Τρίτη, Τετάρτη μπορούμε να κανονίσουμε μια προστή συνειδρίαση, αν θέλετε Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ρωτάει ο Πρόεδρος ο κάθε εισηγητής θα τις έχει τέλος της επόμενης εβδομάδας, Παρασκευή, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, θα έχουμε τις, συμβαστικές, ε, τις πρώτες προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών. Αν χρειάζονται και άλλες προσαρμογές, θα τις κάνουμε τρίτη-τετάρτη. Θα διαπραγματευτούμε μέχρι τέλους. Θα τις έχετε Παρασκευή πρωί. Δεσμεύτηκα ενώπιον των συναδέλφων μου. Παρασκευή πρωί 29 του μήνα. στις 29 εσείς ρωτάει η Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη που επιμένω έτσι 29 στέλνετε τις συμβιβαστικές τροπολογίες ή τις τροπολογίες, συμβιβαστικές τροπολογίες που θα έχετε ξαναδεί με τους διαφορούς σκιώδεις. Θα έχουμε ήδη τις εξετασμένες, αναθεωρημένες ε, συμβαστικές τροπολογίες γιατί ήδη βρίσκονται υπό εξέταση, δηλαδή 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου όλα τα μέλη της Επιτροπής εκτός από τη συνεργασία τους με τους ηγητές, ε, ε, τη συνεργασία με τους ηγητές θα μπορούν να δουν αυτές τις τροπολογίες τέλεια διότι ε, βρισκόμαστε σε επιταχυμένη διαδικασία και πάλι χρειάζεται να έχουμε απόλυτη διαφάνεια ενώπιον των μέλων της Επιτροπής. Θα ψηφίσουμε έτσι λοιπόν από αυτές τις συνθήκες την 5η Ιουλίου. Θα ήθελα να επιθυμίσω όσον αφορά μια δική σας παρατηρήση ότι για την εκθέση του κυρίου Κοζά θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, διότι αυτό το 25% αφορά την εκθέση του κυρίου Κοζά. Σύμφωνο μαζί σας, το μελετώ παράλληλα. Έχουμε τελειώσει με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπούλο για το σχέδιο γνωμοδότησής του για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2013. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα σας δώσω... Εδώ έχουμε μια γνωμοδότηση που αφορά το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013 ε, μετά από τα σχόλια, τη γνωμοδότηση της Κομισιόν. Εγώ χαίρομαι για την αύξηση των πιστώσεων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση των νέων, την διαβίω εκμάθηση σε ένα πλαίσιο και συνθήκες κρίσης όπως χρειάστηκε να αυξήθει αυτός ο προπολογισμό και να υπάρχει ένας προπολογισμό απασχόλησης, όχι λιτότητας αλλά ανάπτυξης της απασχόλησης. Η αύξηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου επιθυμώ τα 22 δισεκατομμύρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα να ανακατανεμηθούν όχι μόνο στις αρχικές χώρες αλλά στο σύνολο των κρατών που θέλουν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των νέων και να υπάρξει μια γρήγορη πολιτική για αυτό το θέμα. Δυστυχώς ε, για το Progress δεν καταφέραμε να αυξήσουμε, έγινε μείωση. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον να είχαμε αυξήσει αυτόν τον προπολογισμό. Προτείνονται δύο πιλωτικά έργα και μία προπαρασκευαστική δράση για την πρόσβαση στην ε, κοινωνική σύγκληση, υποστήριξη των μεταναστών, των απεσπασμένων εργαζομένων και μια πολιτική ένταξη των αστέγων. Υπογραμμίσα επίσης την ανάγκη δημιουργία δέσμευσης ε, για την υποστήριξη της ηθαγένειας μέσω της οποίας το 2013 προωθούμε την ελευθερία κυκλοφορίας, γεγονός που επιτρέπει επίσης ε, απασχόληση και κινητικότητα της απασχόλησης καθώς και το πρόγραμμα νεολαία σε πάντα με το ίδιο σκεπτικό. Αυτές είναι οι κυριότερες μου παρατηρήσεις αναμένοντας το συμβούλιο, τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου στα μέσα Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά, λέει ο Πρόεδρος. Φρέντερικ Νταρντέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω Ε, συμφωνώ γενικά με τον εισηγητή, αλλά έχω τρεις σκέψεις για τρία θέματα. Πρώτα απ' όλα, η αύξηση των πιστώσεων ε, δέσμευσης, ανάληψη υποχρεώσεων ε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είμαι ικανοποιημένο με αυτά και θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη που υπάρχει για τέτοιε πιστώσει για τι πληρώμε. Εγώ, στο πλαίσιο τη εργασία μου στην Επιτροπή Προπολογισμού, διαπιστώσαμε ότι το Συμβούλιο έχει μια τάση να μειώνει αυτέ τι πιστώσει ε, πληρωμή. Ενώ, κατά την απόψη μου, με τον οικονομικό προγραμματισμό τα κατα... λίγουν ε, τα τιμολόγια πρέπει να πληρωθούν και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Η δεύτερη μου σκέψη αφορά την αύξηση των πληρωμών των πιστώσεων ε, για το Ταμείο Προσαρμογής. Είναι σημαντικό. Είναι πεπισμένος ότι πρέπει να επιταχύνουμε, πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επαρκείς πιστώσεις, αλλά προσοχή στους, σε όσους δεν συμφωνούν με το Ταμείο Προσαρμογής. Το είπαμε προηγουμένως, ειδικότερα την εποχή που συζητάμε για τη διατήρηση αυτού του Ταμείου. Τώρα όσον αφορά τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, θα ήθελα να προσθέσω σε όσα ανέφερε ο εισηγητής ε, στην γνωμοδότησή του την προώθηση την, ε, της μετοχικής συμμετοχής των εργαζομένων και στην προπαρασκευαστική δράση για την κοινωνική ένταξη. Το έχουμε ξανααναφέρει που θα επιτρέψει ίσως μια μέρα να ξεκινήσει μια ε, ε, νομοθετική πρωτοβουλία για τα ελάχιστα εισοδήματα. Τέλος, ε, συμφωνώ με την ενίσχυση των πιστοτικών κονδυλίων για την προπαρασκευαστική δράση, όπως αναφέρει ο συγγητής. Θα αποτελέσει μια εγγύηση για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται, επομένως, το λόγο έχει ο εισηγητής. Δεν έχω και πολλά να σας προσθέσω. Πρώτα απ' όλα είπαμε είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Είπαμε για δεν θα υπάρξει πρόβλημα τόσο ώστε να μπορούμε να δούμε σε κάποιο συμβιβασμό. Ε, γιατί είπαμε ότι είναι επίγον κάτι να γίνει όσον αφορά την απασχόληση με την κρίση του χρέους, επομένως θα εξεύρουμε ε, κάποιες λύσεις ε, για το Συμβούλιο και για την Επιτροπή των Προπολογισμών για να είναι σύμφωνοι. Πρόεδρος. Επομένως, προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα καθοριστεί ανάλογα με τι θα γίνει με το κύμα του Συμβουλίου. Για να μπορούμε να έχουμε στην καλύτερη περίπτωση μέχρι τα μέσα Ιουλίου Γιατί είπαμε μέχρι το μεσημέρι της 21ης Αυγούστου και έτσι είναι δυνατόν οι συνάδελφοι ανάλογα με τη θέση του Συμβουλίου να κάνουν τις διακοπές τους και να μπορέσουμε να δούμε θα είναι τις 10 τροπολογίες για να συζητηθούν για να ψηφιστούν στις 6 του μια που το έχουν διάγραμμα δεν και τόσο ευαίσθητο. Τώρα θα φτάνουμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα το πρωί. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μανέσκου για την έκθεσή μας επί της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς για την ιστορική αγορά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο για την αναγκη των οδηγιών ε, κατακύρωσης των δημοσίων συμβάσεων. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στις αναλύσεις που έχουν γίνει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μετά από συναντήσεις διαβούλευσης που είχαμε τα ενδιαφέρομενα μέρη, υπέβαλα 35 τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης που έχω διαβιβάσει και επιθυμούσα να υπογραμμίσω τα ακόλουθα γεγονότα. Η κατοχήρωση δημοσίων συμβάσεων μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ένα εργαλείο χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων του Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία καθώς και την ε, ε, κατοκύρωση δημοσίων συμβασών οικολογικών που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα και να επιτύχουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης. Η στρατηγική 2020 προβλέπει ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να μας επιτρέψουν να ε, ξοδεύουμε καλύτερα τα δημόσια χρήματα υπό τις στρέψεις συνθήκες κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις γίνονται σημαντικότερες από ποτέ. Πρόκειται για ένα εργαλείο κλειδί που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θέσεων εργασίας βιώσιμων που θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θα προωθούν την καινοτομία και την έρευνα και θα ε, στηρίζουν με μία μελιτέο τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει να δώσει τη δυνατότητα επενδύσεων για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Όπως έχω ξαναπεί, οι βιώσιμες θέσεις απασχόλησης αποτελούν έναν από τους μεγάλους στόχους. Το ίδιο και των διακρίσεων και, της κοινωνικής, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θεωρώ λοιπόν η αναθεώρηση της οδηγίας ε, είναι ευπρόσδεκτη, ειδικότερα η οδηγία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Ελπίζουμε ότι οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία θα ενισχυθούν χάρη στην υλοποίηση αυτής της αναθεωρημένης οδηγίας. Τα κόστη που πρέπει να υποστούν οι εταιρείε στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να μειωθούν. Αυτό αποτελεί το αντικείμενο μια από τι τροπολογίε. μου. Λέω ότι αυτά τα κόστη πρέπει να μειωθούν στο μέγιστο χωρί να επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματικότητα. Και σίγουρα χωρί να υποβαθμιστεί η δυνατότητα αυτών των εταιριών να δημιουργούν θέσει εργασία. Χαιρετίζω την πρόταση της Κομισιόν που περιλάμβανε πολλά νέα στοιχεία και που θα καταστήσει αυτή την οδηγία ένα νομοθετικό κείμενο σύγχρονο. Ωστόσο, όλες αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της νομοθετικής απλούστευσης και των κριτηρίων που να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανή, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματικά. Πρέπει επίση να διασφαλίσουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής εκ μέρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσει. να ανατίθενται δηλαδή πολλές συμβάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι έτσι μόνο μπορούν να υπάρξουν βιώσιμες θέσεις εργασίας καλής ποιότητας. Αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων καθώς και τις τροπολογίες τους για αυτό το σχεδίο γνωμοδότησης. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά και να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του συναδελφού Καστέξη που δεν μπόρεσε να παραστεί, έχω να σας πω το εξή για την πολιτική μας ομάδα είναι το θέμα σημαντικό. Γιατί μιλούμε εδώ για χρήση ύδατος, ενέργειας, μεταφορών, ταχυδρομικές υπηρεσίες, που όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι το ελάχιστο το οποίο δίνει ποιότητα ζωής στους λιγότερο πρόμοιους της κοινωνίας. Δεν μπόρεσα τις κυρίες Μανέσκου να αναλύσω όλες τις τροπολογίες, αλλά θα κατεβάσουμε κάποιε τροπολογίες, γιατί εκτό από την αποτελεσματικότητα ε, Έχω, έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ που συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποια μεταβλητή, κάποιο τον παράγοντα δικαιοσύνη. Και αυτά τα βασικά στοιχεία διαβίωσης να συνδέονται από αποτελεσματικότητα, να παρέχονται με ποιότητα σε όλο τον κόσμο. Και πίσω όσον αφορά τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις, θα πρέπει και εδώ να υπάρχει μια κοινωνική πτυχή, αλλά να ληφθεί υπόψη και μεταβλητή τιμή σε σχέση με την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Ποιότητα, δικαιοσύνη επομένω σε αυτή την παροχή των ε, αγαθών δημοσίου ενδιαφέροντος. Πρόεδρος, θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Θέλει μήπως το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια απλή παρατήρηση γενική φύση. Η Κομισιόν ευχαριστεί την Επιτροπή Απασχόληση για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Συμμερίζεται την άποψη της κυρίας Υγεητρίας όσον αφορά της, την ανάγκη διασφαλίσης μια σωστή ισορροπίας αφενός μεταξύ της ανάγκης προώθησης των στόχων του θεματολογίου 2020, δηλαδή καλύτερη κοινωνική ένταξη, προστασία του περιβάλλοντος και κοινοτομία και αφετέρου των αναγκών απλούστευσης των κανόνων, ώστε να μην δημιουργείται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους οικονομικούς φορείς και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, την ανάγκη χρήσης σαφών ενιών ώστε να αποφεύγουμε τις δυσκολίες ερμηνείας και εφαρμογής. Και πάντα να έχουμε υπόψη μας τις αρχές της συνθήκης, τη μη διακριτική μεταχείριση και τη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές που θα θέλουν να μιλήσουν. Όχι κυρία Συγκήτρια. Σας ευχαριστώ, λέει η Γήτρια. Σας ευχαριστώ όλους να αδελφοί όσα είπατε. Και περιμένω να συνεργαστούμε με τους ε, σκιώδες ηγητές για την έκθεση. Θα προσπαθήσω να καλύψω όλες τις απόψεις. την κοινωνική δικαιοσύνη, την εξισορρόπηση μεταξύ των ε, επιμέρους αρχών της ε, στρατηγικής για το 2020, την αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι καταφέραμε να έχουμε ένα πάρα πολύ αξιόλογο έγγραφο τελικά ε, με όλα αυτά σε σχέση με το αρχικό δικό μου κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Τέλεια και τώρα. Με αυτό το σημείο τελειώσαμε για το, για το πρωί. Τέσσερις εβδόμου το μεσημέρι πρώτες μήνες τροπολογίας για να συζητηθούν στις 6 Ενάτου. Τέλος για τώρα το πρωί. Το ραντεβού μας στις 3 η ώρα. Η κυρία Σουέντερ θα προεδρεύσει. Καλό μεσημέρι.